Ladies and gentlemen, good afternoon. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Uh, be welcome uh, to this meeting. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής uh, Νομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με κάποιες αλλαγές που έγιναν στην αρχική ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση των συντονιστών αναβάλλεται για αύριο το πρωί, 9 με 10 παρατέταρτο. Το σημείο 31, με θέμα την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Έντμουντ Στόιμπερ, αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση μετά από έτοιμα του κυρίου Άντερσον των Πρασίνων. Το θέμα της ε, παράληψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε ερώτηση για τη συνθήκη του Μαρακές ε, εμπρόθεσμα και με βάση το κανόνα 130 ε, θα συζητήσουμε για το σημείο αυτό στα διάφορα κατά το τέλος της συνεδρίασης. Ελπίζω να συμφωνείτε με τις προτινόμενες αυτές αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω αντιρρήσεις και ρωτώ αν υπάρχουν ε, άλλες προτάσεις ε, για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω άλλον κανένα. Οπότε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υποβληθούν μέχρι το συνεδρία συνεδρίασης αντιρρήσεις για τα πρακτικά ή διορθώσεις, τα πρακτικά της συνεδρίας 1η και 2 η Δεκεμβρίου ε, του 2014 και της η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2014 θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. 13 και 14. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 Ε, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω την ε, αρμόδια επίτροπο για θέματα δικαιοσύνης ε, καταναλωτών και ισότητας των δύο φύλων, την κυρία Βέρα Γιώραβα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε στην Επιτροπή μας την κυρία Επίτροπο. Θα της δώσουμε το λόγο για μια αρχική παρουσίαση και θα ακολουθήσει γύρω ερωταπαντήσεων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Σφόποντα. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το κοινό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα τόσο νωρί μετά την ανάλυση των καθηκόντων μου. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση προ ε, το το δικό μα όφελο και τη κοινωνία και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προστασία και εμπιστοσύνη για τους καταναλωτές και ευκαιρίες για τις ευκαιρίες. Σε μια δικαιότερη εσωτερική αγορά θα συμβάλλουμε τα μάλα στο να ενισχύσουμε την οικονομική δραστηριότητα, να τονώσουμε την καινοτομία και να εξυγχρονίσουμε την καθημερινότητά μα. Οι τρέχουσες και μελλοντικές μας πρωτοβουλίες θα φέρουν πραγματικά αλλαγές. Και προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αποφασιστικά βήματα. Μάλιστα, η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φερικαιότητα είναι αποφασιστική σημασία. Και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στον εισηγητή τον κύριο Σβιεύκα που εξασφάλισε μια αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων. Γιατί οι έντιμοι επιχειρηματίε αξίζουν βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίε και οι βελτιωμένοι κανόνε για τη δικαιοδοσία θα αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και θα θεσπίσουν κατάλληλα εχέγγυα κατά τη καταχρηστική αναζήτηση τη ευνοϊκότερη νομοθεσία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θέσπιση ενό συστήματος ε, διασυνδεδεμένου μητρώου φερεγγιότητας ή ε, θα διευκολύνει τη διαφάνεια στι διαδικασίε για του ε, για του δανειστέ. Είναι πολύ αυτό το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης και θα δημιουργήσει μια αλλαγή νοοτροπίας στην επιχειρηματική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει όμως να σταματήσουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Μάλιστα, εισακούστηκε το έτοιμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υιοθετήσαμε μία σύσταση για μία νέα προσέγγιση της ε, χρεοκοπίας των επιχειρήσεων. Και μάλιστα μέχρι το Μάρτιο του 2015 θα εφαρμοθεί η σύσταση από τα κράτη-μέλη με η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν και περαιτέρω μέτρα στον τομέα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη πολλά αντικειμενικά εμπόδια που κρατούν ακόμη υποτονική την επιχειρηματικότητα. Μόνο 2% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επενδύουν και σε άλλα κράτη-μέλη, δημιουργώντα ή διηρύοντας οι γιατρικές τους. Μάλιστα, προτείναμε το καθεστώς τη εταιρείας, της ε, ενιαίας σε ένα μέλος για να διευκολυθεί η διασυνοριακή κατάσταση επιχειρήσεων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας, τον κύριο Δεγκράντε Πασκουάλ, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο τομέα αυτό. Μερικοί από εσά εκφράσατε ανησυχίε για το πιθανό αντίκτυπο αυτή τη πρόταση σε διάφορα μοντέλα συμμετοχής των εργαζομένων ή τη αναγκαστική αυτοπασχόλησης. Όλες αυτές οι πτυχέ θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά και να συζητηθούν εκτενώς προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση. Μια πιθανή λύση θα ήταν να θέσουμε την πρόταση στα πλαίσια της ε, ψηφιοποίησης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη ε, διοικητική απλούστευση. Η γενίκευση των ηλεκτρονικών διαδικασιών ε, έχει νόημα στα πλαίσια της προσπάθειας διασυνδεδεμένων μητρών επιχειρήσεων και δυνάμει της αναθεώρησης της οδηγίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και μάλιστα η πρόσφατη οικονομική κρίση προκάλεσε συζήτηση για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Και μάλιστα η σχετική οδηγία για τα ε, δικαιώματα των ε, ιδιοκτητών ε, είναι πολύ σημαντική και ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη για τη συνεργασία που είχαμε. Στη διάρκεια της κρίσης διαπιστώσαμε ότι οι μέτοχοι και ιδιαίτεροι θεσμικοί επενδυτές πολύ συχνά είτε απουσίαζαν είτε, ασκή, είτε ασκούσαν βραχυπρόθεσμη πίεση στις επιχειρήσεις. Έτσι είχαμε ένα κερδοσκοπικό φαύλο κύκλο που διέφυγε του κινδύνου και δημιούργησε πολλά δεινά και αντικσότητες στις κοινωνίες μας. Θέλουμε μια ισορροπημένη λύση μεταξύ των επενδυτών που θέλουν καλύτερη επισκόπηση της κατάστασης και του Διευθυντικού Συμβουλίου που θα πρέπει να κρατήσει τις αρμοδιότητες για σωστή διαχείριση μιας επιχείρησης. Τα θέματα των αμοιβών, των αποδοχών και των συναφών συναλλαγών θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο αυτό. Και μάλιστα ε, οι διάφορε πτυχέ του εταιρικού δικαίου αποτελούν τμήμα μια γενική προσπάθεια για βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και θα ήθελα να σα ζητήσω την υποστήριξή σα και την αθάρισή σα στα θέματα αυτά. Όπω βλέπετε από το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015, η ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι εμβληματική πρωτοβούλια μα βέβαια θα λειτουργήσει μόνο αν αντιμετωπίσουμε και λάβουμε υπόψη τις ανάγκες και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί ακόμη ένα μηδαμινό τμήμα των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών μοντέλων. Μόνο 14% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τις ε, πωλήσει μέσω διαδικτύου και μόνο 5% των επιχειρήσεων έχουν διασυνοριακές πωλήσει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όμως αναπτύσσεται ραγδαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετησίω ε, το ποσοστό ανάπτυξης του είναι 10%. Οι καταναλωτές ε, δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην ε, διασυνοριακή αγορά άλλων χωρών. Προτιμούν την, διασυνορι... την ηλεκτρονική αγορά στην ντόπια, τις ηλεκτρονικές αγορές στις ντόπιες αγορές και μάλιστα ένα κοινό, είναι σημαντικό να έχουμε ένα κοινό δίκαιο για τις πωλήσει που θα περιλαμβάνει και τις ηλεκτρονικές πωλήσει. Βέβαια, η σχετική πρόταση δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει απαραίτητη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Θέλουμε να την αποσύρουμε λοιπόν και να υποβάλουμε μια τροποποιημένη πρόταση φέτος για τον ενιαίο νόμο και το δίκαιο για τις πωλήσει. Και μάλιστα θα είναι μια από τις νέες πρωτοβουλίες του πακέτου μας για την ενιαία ψηφιακή αγορά θέλουμε να δούμε ποια είναι τα εμπόδια στο ενιαίο ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο. Και στη διαβούλευση αυτή θα ήθελα να αξιοποιήσω και τις δικές μας συζητήσεις ε, για να βελτιωθεί το κοινό δίκαιο πολίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για την αγορά ψηφιακών προϊόντων και τα βασικά δικαιώματα για προϊόντα όπως ε, ε, ε, αθλητικές, ε, αναμετάδοση αθλητικών ε, εκδηλώσεων ή μουσικών κομματιών δεν, είναι, δεν ρυθμίζονται επαρκώς. Θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί με εμπιστοσύνη να αγοράζει ηλεκτρονικά και σε άλλες χώρες μέλη με την ίδια ευκολία που το πραγματοποιεί και στην πατρίδα του και να αναζητά τα καλύτερα προϊόντα, τα πιο ποιοτικά και στις φθηνότερες τιμές. Και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους χωρίς περιττό κόστος και μάλιστα κάποιος ε, Ούγγρος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα βρετανικό ε, ιστότοπο τα αγαπη, τους αγαπημένους του αγώνες και ο ένας πάροχος θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει ελεύθερα τις, τις υπηρεσίες του σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο πολιτικό μείγμα και να αντιμετωπίσουμε την, τον νομικό κατακαιρματισμό που υπάρχει στην ψηφιακή αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστή προστασία των καταναλωτών. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να συνεργαστούμε στενά, έχοντα υπόψη ότι όποια πορεία και αν ακολουθήσουμε, θέλουμε μία λύση που να συνάδει με την, κοινωτική, την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Θα ήθελα όμως να ολοκληρώσουμε και άλλα δύο θέματα για να διευκολύνουμε τους Ευρωπαί... Ευρωπαίους πολίτες να διαμένουν και να ταξιδεύουν στο εξωτερικό τα σύμφωνα συμβίωσης, οι γαμικές σχέσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία αγορά για να μειώσουμε το άχθος για τους πολίτες. Και να, οι διαδικασίες να μην είναι χρονοβόρες ούτε ακριβές. Βασίζομαι σε εσά για να λάβω την υποστήριξή σας για αυτά τα δύο θέματα και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε επιτυχές αποτέλεσμα. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσω ένα ανοιχτό διάλογο μαζί σας, χωρίς ταμπού, σε ό,τι αφορά το, τη μελλοντική μας ατζέντα, τα μελλοντικά μας θέματα. Ας μιλήσουμε για το οικογενειακό δίκαιο. Το 2015 σκοπεύω να εστιάσω στην αναθεώρηση της λεγόμενης ε, του καονισμού 2A ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα γαμικού δικαίου και γονικής ευθύνης. Στο παρελθόν, στο παρελθόν οι διαφορές εντός οικογένειας έχουν αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μεγαλύτερης κινητικότητας των πολιτών. Τον Απρίλιο του 2014 ε, η Κομισιόν έκανε μία διαβούλευση που δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε στοχευμένες βελτιώσεις στους κανόνες ε, που ισχύουν. Χρειαζόμαστε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς να δούμε ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο, να αναγνωριστούν οι αποφάσεις και να εφαρμοστούν σε διασυνοριακές καταστάσεις. Θα κάνω λοιπόν μια πρόταση ακριβώς γι' αυτό. Η αυξανόμενη κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σημαίνει ότι έχουν, έχουμε και πιο συχνές σχέσεις με άλλους πολίτες και με τρίτες χώρες ε, και με επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Επομένως, οι διεθνείς συμφωνίες είναι απαραίτητες για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου θέλω να ενισχύσω την πολυμερή συνεργασία στον εξαιτορικό τομέα της αστικής δικαιοσύνης. Σκοπεύω λοιπόν να συμμετάσχω ενεργά στην δουλειά που θα κάνει ε, η διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, όπου θα συμμετάσχουν οι πιο μεγάλες οργανώσεις στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, όπου εμείς είμαστε μέλους από το 2007. Ο σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεών μας πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, η Κομισιόν προτείνει την προσχώρηση σε σχετικές διεθνείς συμβάσεις, όπως παραδείγματο χάρη η Σύμβαση της Χάγης του 1988 για την διεθνή απαγωγή. Είναι ένα βασικό εργαλείο Υπάρχουν 93 συμβαλόμενα μέρη και η Σύμβαση του 96 για την προστασία του παιδιού. Πολύ πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απαγωγής των παιδιών συμπεριλαμβάνει την αποδοχή της προσχώρησης τρίτων χωρών στην Σύμβαση του 1988. Όμως η, προσπάθ... η άσκηση αποκλειστικής αρμοδιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα, όπου απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Θέλω μαζί με τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουμε έντονο συντονισμό και γρήγορη συμφωνία για τι μελλοντικέ προσχώρήσει. Η Κομισιόν πρότεινε, όπω ξέρετε, να δεχτούμε την προσχώρηση 8, τρίτων, 8 νέων τρίτων χωρών στην Σύμβαση για την Απαγωγή του Παιδιού. Η Κομισιόν ε, υποστηρίζει στενά αυτές, θερμά αυτές τις προτάσεις και ελπίζω ότι το θέμα της αρμοδιότητας έχει ξεκαθαριστεί από το δικαστήριο. Και επομένως μπορούμε να περάσουμε σε μια γρήγορη συμφωνία στο Συμβούλιο για το αστικό και εμπορικό δίκαιο. Η Κομισιόν ασχολείται σε προπαρασκευαστικό στάδιο ε, στις εργασίες που γίνεται στην ε, Χάγη για να υπάρξει μια ευρεία ε, σύμβαση για την εκτέλεση των αποφάσεων, η λεγόμενη, ε, το λεγόμενο σχέδιο περί αποφάσεων. Μια διεθνή σύμβαση για αυτό το θέμα θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στη νομική προστασία των εταιριών μας και των πολιτών μας ε, παγκοσμίω. Θα δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εμπορεύονται στο εξωτερικό και οι πολίτες να ταξιδεύουν παγκόσμια σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Εντάσσεται ωραία στην ε, εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται πολύ τεχνικά, αλλά ο τελικός στόχος είναι απλός. Η ζωή των πολιτών μας να γίνει πιο απλή, με αυτό το στόχο κατά νου δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις προτάσεις που υπάρχουν ήδη επιτάπητος. Να μιλήσω για δύο προτάσεις πιο συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του καονισμού που καθορίζει μια ευρωπαϊκή διαδικασία για τις μικρές απαιτήσει, μικρές αξιώσεις. Ε, θα ξέρετε την προσέγγιση του Συμβουλίου. Η Κομισιόν παραμένει πεπισμένη ότι αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κατόφλι που έχουμε μέχρι στιγμής ε, στα 2.000 ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί. Γιατί οι διασυνοριακές απαιτήσει συνήθως εντός της Ευρώπης είναι περίπου 40.000 ε, ευρώ στην Ευρώπη. Ο κύριος Τεμπεργκ είναι εισηγητής και ξέρω ότι αν έχουμε ε, αποτελεσματικά ένδικα μέσα, είναι αυτό ένα φράγμα για την απάτη Σε ό,τι αφορά την απλούστευση της αποδοχής κάποιων δημοσίων εγγράφων, ε, χαίρομαι που στήριξε το Κοινοβούλιο τη δική μας πρόταση το Συμβούλιο. Γενικά συμφωνεί με τους στόχους απλούστευσης της πρότασης, αλλά αμφισβητεί το πεδίο εφαρμογή. Είμαι πεπισμένη ότι όταν ρυθμιστεί το θέμα του πεδίου εφαρμογή, όλα τα υπόλοιπα ε, θα ρυθμιστούν. Α συνεργαστούμε ούτω ώστε να βρούμε κοινό έδαφο, ούτω ώστε και οι πολίτε και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις δαπανηρές και γραφειοκρατικές διατυπώσεις των συντομότερων δυνατών. Θα ήθελα, εν κατακλείδη, να μιλήσω για το πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη και τη σημασία του. Ε, ετοιμάζουμε τώρα την τρίτη εκδοχή αυτού του πίνακα. Ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα είναι ο πυρήνας της ε, κοινωνίας και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη. Θέλω να συνεργαστούμε τόσο ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτό το εργαλείο. Μηχανισμοί επίλυση των διαφορών. Οι μηχανισμοί αυτοί θα παίξουν σημαντικό ρόλο στα δικαστικά συστήματα και ο επιγραμμικός, η επιγραμμική επίλυση των διαφορών που θα είναι λειτουργική το 2016 το διαδίκτυο θα είναι επιπλέον χρήσιμο εργαλείο. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω ότι ο εναλλακτικός, η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών θα πρέπει να ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία των κρατών μελών φέτο. Θα είναι απλό, αποτελεσματικό, γρήγορο, φθηνό εργαλείο για να επιληθούν διαφορές εκτός δικαστηρίου σε διαφορές καταναλωτών. Θα υποφευθούν και οι καταναλωτές και οι έμποροι, γιατί θα αποφευθούν οι δαπανηρές και χρονοβόρε ε, διαδικασίες στο δικαστήριο. Έχουμε αυτές τις τεχνικές λοιπόν εξελίξεις στις 25 και 27 έως 27 Νοεμβρίου του 2014 η Κομισιόν έκανε ε, ένα τεστ ενός πρωτοτύπου με 120 συμμετέχοντες και μια έκθεση για τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο την Άνοιξη. Τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό ε, νομικό πλαίσιο ε, για να βοηθήσουμε την κατάρτιση των επαγγελματιών της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να με υποστηρίξετε θερμά γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, I Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τις ε, αρχικές σας παρατηρήσεις. Μας δείξατε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, το πρόγραμμά σας αλλά επίσης και το ότι αντιληφθήκατε το ερώτημα που ετέθη στην πρώτη ακρόαση του Κοινοβουλίου πριν αναλάβετε τα καθηκόντά σας. Είστε θα έλεγα η, επιτροπή που, η Επίτροπος που είναι πιο κοντά στην Επιτροπή μας και είμαι σίγουρος τώρα πως οι βουλευτές ε, θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να κάνουμε έναν ε, πραγματικό διάλογο ο οποίος ε, θα προωθήσει το κοινό μας πρόγραμμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, βουλευτές να τηρήσουν τον ε, χρόνο. Λοιπόν, έχουμε ήδη τον καταγωγητή, ο κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγες μέρες ε, εγκρίθηκε ο κανονισμός για τις διασυνοριακές αποφάσεις ο κανονισμός Βρυξέλλες 1. Αλλά βεβαίως ξέρετε πως εξαρτάται από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, πως θα μπορεί να ξέρει ένας δικαστής ότι έγιναν σεβαστά τα δικονομικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων, ειδικά όσον αφορά τα εντάλματα, τη συλλογή δεδομένων ε, και τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Είπατε πως ε, θα εργαστείτε προς κάποιες ε, ελάχιστες δικονομικές εγγυήσεις ε, για να υπάρξει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων δικαιοσύνης. Ε, πώς προχωράει αυτό το ζήτημα και πότε θα μπορούμε να περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Η επόμενη ερώτησή μου αφορά την πιθανή κωδικοποίηση οδηγιών για το εταιρικό δίκαιο, το πρόγραμμα εργασίας του 2015, κάτι το οποίο σημαίνει πως πρέπει να αναμένουμε σύντομα κάποια αποτελέσματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αυτό το θέμα. Αν μου επιτρέπετε. Θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, ζητήθηκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά και να ευχαριστήσω εγκάρδια την ε, κυρία Επίτροπο για την ε, ενημέρωση που έκανε. Λυπούμε που δεν ήμουν από την αρχή, αλλά με τις αεροπορικές συνδέσεις, ιδιαίτερα Δευτέρα, είχα πρόβλημα, πρόβλημα με το να φτάσω έγκαιρος. Και τα σχέδια και οι πρωτοβουλία σας ε, συνάδουν με τις δικές μας προσδοκίες και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί συμπεριλάβατε όλα αυτά τα θέματα και μάλιστα ως προτεραιότητες στο πρόγραμμα εργασιών σας για το 2015. Ε, ιδιαίτερα η αναθεώρηση της οδηγίας και του κανονισμού Βρυξέλλας 2. Ο κανονισμός αυτός αφορά θέματα που επηρεάζουν πραγματικά την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών ιδιαίτερα όταν αλλάζει το προσωπικό καθεστώς, όταν γίνονται κάποιοι μεικτοί γάμοι, όταν αλλάζει κανείς ε, τόπο διαμονής. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την οικογενειακή ασφάλεια και κυρίως την ασφάλεια των παιδιών, γιατί είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες και θα πρέπει να προστατευτεί σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς αυτή η ασφάλεια. Οπότε είναι σημαντική η αναθεώρηση αυτού του κανονισμού και καλό θα ήταν να επιταχυνθεί αυτή η αναθεώρηση και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη 14η οδηγία για τα δικαιώματα των εταιριών και κυρίως ε, την ε, διασυνοριακή, τη μεταφορά ε, διασυνοριακά της έδρας. Το 2012 ε, υιοθετήσαμε μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, με αυτό ακριβώς το αντικείμενο και νομίζω ότι από κάθε άποψη θα ήταν θετική η ανάληψη και νομοθετικής πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Χαίρομαι επίσης ε, για την πρόθεσή σας να ασχοληθείτε το συντομότερο δυνατό με τη συνέχεια του σχεδίου Justice Scoreboards, του πίνακα αποτελεσμάτων δηλαδή για τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση ε, να μην ξεχάσετε αυτό το θέμα και στις συναντήσεις που θα έχετε με τους υπόλοιπους επιτρόπους ε, να φροντίσετε ώστε ο πίνακας αποτελεσμάτων ε, να αξιοποιηθεί για να έχουμε έμπρακτη βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης στις διάφορες χώρες μέλη. Και να μην ε, ε, γίνουν κάποιες πολιτικές προσπάθειες ε, για μη σωστή αξιοποίηση του πίνακα αυτού αποτελεσμάτων. Είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου αλλά και για θέματα ποινικού δικαίου. Απευθύνω έκκληση λοιπόν να υιοθετήσετε στεναρή θέση σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια έγγραφα. Δεν ξέρω αν ήδη αποφασίσατε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν οι σχετικές εργασίες σας. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ε, καταλήξαμε σε ε, ένα σημαντικό αίτημα. Δεν αρκεί η προσπάθεια, μάλλον δεν έχει νόημα ξεκέλευθων αλλαγών. Γιατί πραγματικά η πάλι κατά της γραφειοκρατίας είναι ε, από τις σημαντικότερες μάχες που έχουμε να δώσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά αντί να έχουμε επαναστατικές ε, μεθόδους, καλύτερα να έχουμε μια σταδιακή και βήμα προς βήμα ρυθμίση. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από τα απλά πράγματα και να ασχοληθούμε μετά με τα πιο περίπλοκα. Δηλαδή να μην γίνουν αυθείς αμέσω κάποιες επαναστατικές αλλαγές, αλλά σταδιακές μικρές αλλαγές. Το συντομότερο όμω δυνατό να τεθούν σε εφαρμογή. Επίσης, ο συνάδελφο μίλησε για τον κανονισμό Βρυξέλλες 1. Απασχόλησε τη νομική επιτροπή για πολλά χρόνια. Είναι σημαντική η εμπιστοσύνη του πολίτη στην απονομή δικαιοσύνη και στο δικαιικό σύστημα τη κάθε χώρα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Και επίσης πρέπει να στηρίξουμε τα εθνικά όργανα απονομή τη δικαιοσύνης, ώστε να ενστεριστούμε τον καλύτερο τρόπο και να εφαρμόσουν τι ε, κοινοτικέ ρυθμίσει. Και επίση αυτό θα πρέπει να γίνεται με έντιμο τρόπο και με καλή βούληση συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία. Γιατί αυτό το νόημα έχουν και οι αλλαγές ε, στον κανονισμό Βρυξέλλες 1. Και ελπίζω ότι όλοι αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν. Τέλος, για τις μικροδιαφορές, τα small claims. Ε, φυσικά συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να βρούμε το σωστό ύψος, αν θα είναι 5.000 το ύψος του ποσού, αν θα είναι 5.000, 10.000, 8.000, 15.000 ευρώ, ποιο θα είναι το κατόφλι για να χαρακτηρίζονται μικροδιαφορές. Ε, σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλό το ποσό αυτό. Γιατί θέλουμε η διαδικασία για τις μικροδιαφορές να γίνει ένα πραγματικά εύχριστο εργαλείο νομικό. Θα ήθελα και πάλι να σε ευχαριστώ και να σε ευχηθώ καλή επιτυχία στην υλοποίηση των σχεδίων σας για το 2015. Take a third. Ε, ωραία, θα ακούσουμε τώρα και άλλες ερωτήσεις από την κυρία Χάουτελα και θα περάσουμε στις απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Σας διαβεβαιώ πως η Επιτροπή μας ε, μάλλον θα δώσει θετική ψήφο όσον αφορά στις 8 εκθέσεις για την ένταξη τρίτων χωρών στην ε, Σύμβαση της Χάγης για την απαγωγή παιδιών του 1980 και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει θα γίνει γρήγορα στα άλλα θεσμικά όργανα. Τώρα, είπατε πως ε, θέλετε να συνεργαστούμε σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, σύμφωνα συμβίεσης ε, κτλ. Ποιο είναι το όραμά σας, ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για το ότι πολλά κράτη-μέλη ήδη αναγνωρίζουν κάποια σύμφωνα συμβίωσης. Πού πάμε λοιπόν και πόσο αισιόδοξοι είστε για το ότι θα καταλήξουμε σε μια πρόταση και μια απόφαση. Τώρα να έρθω σε κάτι διαφορετικό. Οι γυναίκες στα ΔΣ εταιριών υποθέτω πως εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε για αυτή την πρόταση. Το συζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο, αλλά θέλω να ακούσω από εσά τι θα κάνετε. Ε, υποθέτω πως ε, υπάρχουν περιπτώσεις ε, που αποδεικνύουν πως πρέπει να γίνουν κάποιες θετικές διακρίσεις. Και για να φύγουμε από τον σκανδαλωδός χαμηλό αριθμό γυναικών στα ΔΣ και αυτό βέβαια πρέπει να πάει μαζί με τις προσπάθειες για να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις για να υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων από το οποίο να μπορούν να επιλεχθούν για το ΔΣ. Thank you for, all the questions. Perhaps... Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Ξέχασα να πω κάτι στην αρχική μου παρέμβαση, πως βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και σε άτυπη βάση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις επίσημες ε, συναντήσεις μας. Όποτε έχετε κάποιες ερωτήσεις μπορείτε να έρθετε σε επαφή ε, μαζί μου. Όσον αφορά τώρα τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, ε, υπάρχει μια πρόταση που είναι μια αντίδραση στον σκανδαλωδώς ε, χαμηλό αριθμό γυναικών στα ΔΣ εταιριών. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, κυμαίνεται γύρω στο 16%. Στη χώρα μου είναι γύρω στο 10%. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εγώ είμαι υπέρ της πρότασης γιατί δεν είναι μόνο δίκαιο να βοηθήσουμε τις γυναίκες, αλλά το να προωθήσουμε κάτι τέτοιο σημαίνει πως προωθούμε την οικονομία, γιατί η ποικιλομορφία ε, είναι βεβαίως ένα πλεονέκτημα και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Είχα εγώ μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με επικεφαλής εταιριών στην Τσεχία και είπαν όλοι πως ψάχνουν γυναίκες γιατί δεν θέλουν να πάει χαμένο το ταλέντο που υπάρχει. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλουμε οπωσδήποτε να προωθήσουμε. Πολλά κράτη-μέλη πρέπει ε, να ενταχθούν και να συμφωνήσουν με αυτή την προσπάθεια. Θα πιέσω οπωσδήποτε για αλλαγή σε πολλά κράτη-μέλη τις επόμενες ε, εβδομάδες. Τώρα για σύμφωνα συμβίωσης ε, και το οικογενειακό δίκαιο Εκκρεμεί εδώ πέρα νομοθεσία. Μίλησα με τον Πολωνό Υπουργό για τη θέση της ε, Πολωνίας ε, και μιλήσαμε και με την ε, Λετωνική Προεδρία για τα κοινά αποκτήματα στον γάμο. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν με κάποια κράτη-μέλη που πρέπει να αλλάξουν την θέση τους επί της προτάσεως αυτής και να γίνει και μια πρόταση και για το σύμφωνο συμβίωσης ε, καθ' αυτό. Οπότε φαντάζομαι πως ε, στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θα επανέλθει αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο. Αισιόδοξα το λέω αυτό. Γιατί έτσι ε, θα βοηθήσουμε και τα παντρεμένα ζευγάρια και αυτούς που έχουν σύμφωνο συμβίωσης για τα προβλήματά τους όταν ε, ταξιδεύουν και ζουν ε, στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα τις ε, μικροδιαφορές, είναι προφανές ότι έτσι θα βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είμαι σίγουροι ότι τους επόμενους έξι μήνες θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για το όριο γιατί όλα τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της νομοθεσίας και οπωσδήποτε υπάρχει βούληση για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θέλω τώρα να κάνω κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι αυτό το όριο. Αλλά θα το διαπραγματευτούμε οπωσδήποτε έντονα συμφωνώ πλήρως τώρα πως η επιβολή του, των Βρυξελών 1 είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή είναι και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που μου κάνατε. Γιατί ο κανονισμός αυτός ε, δίνει μια ε, νομική βεβαιότητα για το θέμα της ε, δικαιοδοσίας ε, των δικαστηρίων ε, και της εφαρμογής ε, των αποφάσεων. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να υπάρξει κάποια εμπιστοσύνη και βεβαίως αυτό σημαίνει πως πρέπει να βασιζόμαστε σε περισσότερη ακριβώς αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο κανονισμός λοιπόν και ελπίζουμε πως η επιτυχής εφαρμογή του θα μας οδηγήσει σε κάποια πρόοδο. Για να μειώσουμε την γραφειοκρατία και τα εμπόδια για τους πολίτες ε, ε, που ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τα δημόσια έγγραφα. Αντιλαμβάνομαι τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των εγγράφων που θα αναγνωρίζονται διασυνοριακά όμως η θέση του Συμβουλίου ήταν να μειωθεί ο αριθμός τους, οπότε θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω λοιπόν πως σε έξι μήνες επιλετονικής Προεδρίας θα καταλήξουμε για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος για μια συμβιβαστική θέση για τον πίνακα βαθμολογίας ε, της δικαιοσύνης. Ε, ε, εκτιμώ περισσότερο αυτό το μέσο όσο περνάει ο καιρός γιατί μας δίνει μια εικόνα της κατάστασης στα κράτη-μέλη στις διαδικασίες αστικού δικαίου μας δίνει την εικόνα αποτελεσματικότητας ε, της ε, δικαιοσύνης ε, και βεβαίως θα το χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο με τον καλύτερο τρόπο για να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη εκεί όπου υπάρχουν κενά να κάνουν κάποια πραγματικά βήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση γνωρίζετε πως ε, ξέρετε, από καιρού καιρών υπάρχει και διεύρυνση, υπάρχει πρόταση για διεύρυνση του πίνακα αυτού και στις ποινικές διαδικασίες. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος να το διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη για να καλυφθεί και αυτό. Αλλά ε, εγώ το θεωρώ χρήσιμο και αναγκαίο να δούμε και την κατάσταση στην ποινική δικαιοσύνη. Τώρα για τις Βρυξέλλες 2α. Το ερώτημα ήταν αν θέλουμε να τον αλλάξουμε και να τον ενημερώσουμε. Τον κανονισμό να σας ενημερώσω λοιπόν πώς θα θέλαμε να δώσουμε την δυνατότητα στους συζύγους να διαλέγουν το δικαστήριο το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη διάσταση ή το διαζύγιο τους, ε, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα βεβαίως μιας φιλικής λύσης όπου αυτό είναι δυνατόν και βεβαίως είναι πάντα προς το συμφέρον των παιδιών, κάτι το οποίο είναι η προτεραιότητά μας. Θέλουμε επίσης να διευκολύνουμε να μπορούν οι οικογένειες να απευθύνονται σε μία μόνο υπηρεσία να υπάρξει δηλαδή μια ενοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών αυτών, ε, διαζυγίου, διάστασης, ε, το ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ε, τα ιστορικά στοιχεία μετά να καταργηθεί καταργηθεί το εκτελεστήριο όσον αφορά τα τις υποθέσεις που αφορούν τα παιδιά, ακριβώ για να μην καθυστερούν, να τεθούν επίσης ε, κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλα τα κρατη να απλοποιηθεί και να ξεκαθαρίσει η διαδικασία επιστροφής ε, παιδιών που έχουν απαχθεί ακριβώς για να μην βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον. Ε, τέλος, να τεθούν κάποιες προδιαγραφές ε, για την επιβολή αυτών των αποφάσεων και τέλος ε, να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και της ε, κοινωνικής πρόνοιας και άλλων αναλόγων υπηρεσιών για να προστατευτούν τα συμφέροντα του παιδιού. Αυτά είναι τα βασικά. Ε, ε, έχουμε ακόμα πέντε ευρωβουλευτές που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Και έχουμε και τον κύριο Τίμερμανς που περιμένει έξω από την αίθουσα. Να ζητήσω από τους βουλευτές να κάνουν σύντομα τις ερωτήσεις τους. Και η Επίτροπος σύντομα να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Είναι η πρώτη συνάντησή μας, ούτως ή θα έχουμε και άλλες στο μέλλον. Κυρία Κούτερλαντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιούροβα για την παρουσίασή σας και για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας. Είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Η ερώτηση. για την πρόταση για τις εταιρείε. Το συζητήσατε, δεν το κατάλαβα ακριβώς το θέμα. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε. Κάποια τμήματα των προτάσεων για αυτές τις εταιρείε θα τα πάρετε και θα τα βάλετε σε άλλα νομοθετήματα. Άρα θα αποσυρθούν αυτές οι προτάσεις ή θα γίνει το σχετικό νομοθέτημα πιο ισχυρό, ούτω ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουν το, αυτά τα στοιχεία οι εταιρείε, ούτω ώστε να παρακάμψουν την φορολογική νομοθεσία. Ίσως θα επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας έτσι. Ε, έχουμε διάφορες ε, ανησυχίες ε, για το θέμα αυτό. Τελικά θα πάρετε στοιχεία αυτού του νομοθετήματος και θα εντάξετε σε άλλες ε, οδηγίες ή κανονισμού, σε άλλα νομοθετήματα. ούτω ώστε να μην χρησιμοποιούν με λαθασμένο τρόπο την νομοθεσία οι εταιρείε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιούροβα για αυτά τα οποία μας είπατε. Τρία ερωτήματα θα ήθελα εγώ να κάνω. Πρώτον, θεωρώ πως ε, δεν μπορούμε μετά τα όσα έγιναν στο Παρίσι να περνάμε απλά στην ημερήσια διάταξη. Για μένα είναι σημαντικό ποια είναι η θέση σας στη σχέση περιορισμού των ελευθεριών και ασφάλειας. Υπάρχει μια συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη Γερμανία υπάρχει συζήτηση για την αποθήκευση δεδομένων, για τα δεδομένα αεροπορικών επιβατών και θέλω να μάθω πώς εσείς ως αρμόδια επίτροπος ε, για νομικές υποθέσεις ε, βλέπετε τη σχέση μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Δεύτερον, έχουμε τις ατομικές ε, εταιρείες. Εκεί πέρα θεωρούν πως επηρεάζονται και κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, δεν θα προωθήσει τίποτα θετικό αυτό στην Ευρώπη. Τρίτον, για, το ψηφια... για την ψηφιοποίηση της Ευρώπης υπάρχει η τεράστια ανασφάλεια των ε, καταναλωτών ε, για την παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπουντά. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο που βρήκε χρόνο στο γεμάτο χρονοδιάγραμμά της ε, για να έρθει και να μας δώσει κάποιες απαντήσεις και στοιχεία. Ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αφορά την αφαιρεγκαιότητα και τη στάση πληρωμών φυσικών προσώπων. Γιατί πολλοί δυστυχώς συμπολίτε μας κάποια στιγμή δεν μπορούν να πληρώσουν, να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τι νομικό πλαίσιο θα προτείνετε για την κατάσταση αυτή, γιατί με την τρέχουσα κατάσταση έχουμε μεγάλη αδικία και ανισορροπία μεταξύ της ρύθμισης που ισχύει για τις ε, αφαιρέγγες επιχειρήσεις και τη ρύθμιση που ισχύει για τους αφαιρέγγιους ιδιώτες. Επίσης, τι γίνεται με την γνωστή και διαβόητη δικτατορία των τραπεζών. Πολλά είναι τα θύματα αυτού του καθεστώτος και πολλοί άνθρωποι εξαιτία ε, της ε, οικονομικής τους ε, ανέχειας δεν μπορούν να αποπληρώσουν ε, τις δόσεις στεγαστικών δανείων, για παράδειγμα, και χάνουν τα σπίτια τους. Άλλο πρόβλημα που έχουμε στη Ρουμανία είναι η, τα στεγαστικά δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου εξαιτία ε, της αύξησης της τιμής του φράγκου και της ανατροπής αυτής της συναλλαγματικής ισοτιμίας σχέση με το ευρώ, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε δινή κατάσταση. Τι θα προτείνετε θα υιοθετήσει το γαλλικό μοντέλο που ισχύει και σε άλλες νομικές ε, καταστάσεις και ένομες τάξεις. Ευχαριστώ. Η νέα Επιτροπή σημειώνει μια πολιτική ασυνέχεια σε σχέση με τις δεσμές που είχε αναλάβει η προηγούμενη. Η Κομισιόν αποφάσισε να αποσύρει τις, ε, κάποιες προτάσεις που δεν έχουν ε, καταλήξει, ας πούμε, και που δεν έχουν μέλλον και θα εστιαστεί, υποτίθεται, στα σημαντικά. Έχετε πάρει λοιπόν μια πολιτική δέσμευση. Γι' αυτό στην ε, λίστα των προτάσεων που θα αποσυρθούν, ε, αν δεν υπάρξει συμφωνία, έχετε την οδηγία για την ε, μητρική άδεια. Γιατί υπήρξε αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Γιατί δεν προστατεύονται έτσι οι μητέρε εργαζόμενοι και τα παιδιά του. Και ένα άλλο λόγο είναι γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλε τι εργαζόμενε με ισότιμο τρόπο. Πώ θα ξεπεράσει η Κομισιόν αυτό το πρόβλημα, τι πληροφορίε μπορείτε να μα δώσετε για αυτή την πρόταση οδηγία που. Τη νέα, μια ίσως νέα πρόταση η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτή η οποία δεν τελεσφόρησε στο Συμβούλιο. Τελευταία ερώτηση. Η κυρία Ροζιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Θα σας να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Γρήγορα να μιλήσω για κάποια θέματα που ακούστηκαν. Το πρώτο είναι το ευρωπαϊκό δικαίωμα πώληση. Είπατε ότι η πρόταση θα ξαναπροταθεί με κάποιες αλλαγές. Ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της νέας πρότασης. Θα υπάρχει και ένα το καθεστώς ή θα κάνουμε μία μέγιστη ή ελάχιστη εναρμόνιση. Ποια θα είναι η φιλοσοφία της νέας πρότασης. Επίσης, είπατε κάτι για την ε, διάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου στην ευρωπαϊκή αγορά. Όταν έχουμε πρόσβαση σε ένα περιεχόμενο, ε, το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε στην χώρα της συνήθους κατοικίας δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόσκομα. Όμως αν έχουμε μόνο ευρωπαϊκές άδειε μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες σε όλους αυτούς που διαδίδουν περιεχόμενο και που είναι εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο και μπορούσαν να εγκαταστηθούν σε μια χώρα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες όμως. Έχετε μελετήσει την επίπτωση που θα έχει η πρότασή σας και πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτοί που διαδίδουν περιεχόμενο να διαδίδουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο που το θέλουν καταναλωτές. Υποστηρίζεται επίσης την πρόταση ισότιμης εκπροσώπης ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιριών. Χαίρομαι. Για τα δικαιώματα των γυναικών όμως ε, υπάρχει το πρόβλημα του κειμένου για την ε, μητρική άδεια. Ε, πώς θα εξακολουθήσει η γυναίκα να έχει την σωστή θέση, τη θέση που της αρμόζει στον οικονομικό βίο, αν δεν προωθηθήσετε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, η Επίτροπος θα ήθελα να, θα ήθελα να απαντήσει μόνο στις ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Εντόπισα τουλάχιστον δύο ερωτήσεις οι οποίες εκφεύγουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Δεν θα τις απαντήσει η Επίτροπος. Η Επίτροπος έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα δώσω τις απαντήσεις στα τσεχικά, γιατί μπορώ να μιλώ πιο γρήγορα τη μητρική μου γλώσσα και νιώθουμε και αυτή την πίεση χρόνου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άδεια το θέμα αυτό δεν θα το σχολιάσω τώρα. θα πρέπει να προβλέψουμε ένα εξάμεινο χρονικό διάστημα για να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν τη θέση τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τις πωλήσει, αναλύουμε τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών. Έχουμε μια συμβουλευτική ομάδα που εξετάζει όλες τις ε, πιθανότητες και θα δούμε αν μπορέσουμε να επιτύχουμε μια εναρμόνιση και ένα 21 29ο καθεστώς, ένα ευρωπαϊκό δηλαδή καθεστώς που θα διέπει το δίκαιο για τις πωλήσει και που θα ε, ισχύει έναντι των 28 χωρών μελών. Σε ό,τι αφορά τη ψηφιακή αγορά, στα τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε ε, και θα υποβάλουμε τη σχετική πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ισορροπία που θα πρέπει να βρεθεί μεταξύ των ελευθεριών και της δικαιοσύνης, αυτό είναι μάλλον θέμα και αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά είναι ακριβώς επίκαιρο το θέμα και θα φροντίσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και δικαιωμάτων. Θα συνεργαστώ για το θέμα αυτό με τους ε, άλλους επιτρόπους. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία γενικώ των συμπολιτών μας. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και να μην εθετήσουμε δυσανάλογη αντίδραση και μέτρα μετά τα επεισόδια που έγιναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δικαιώματα δημιουργού, πνευματικά δικαιώματα και συναφή ή το θέμα του single member company. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ε, για να καταλήξουμε σε μία πρόταση. Και πάλι θα, θα πρέπει να βρούμε εδώ τη σωστή ισορροπία για να αποφύγουμε κατάχρηση αυτού του μοντέλου, ε, κοινού μοντέλου ε, εταιρεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αφαιρεγκαιότητα, τέθηκαν δύο ερωτήσει σχετικά. Θα εξετάσουμε το θέμα ιδιαίτερα της αφαιρεγγιότητας των φυσικών προσώπων που μερικές φορές ε, υφίστανται τη δικτατορία των τραπεζών και των τραπεζιτών. Θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για τα φυσικά πρόσωπα και τι μέτρα μπορούμε να θεσπίσουμε ή να προτείνουμε ένα κανονισμό που να διέπει την ε, αφαιρεγκαιότητα και την ρυθμίση αυτή με διασυνοριακό τρόπο. Θα πρέπει όμως να γίνει προηγουμένως μια αξιολόγηση της κατάστασης. Ευχαριστώ θερμά όλους σας για τις ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη αν δεν έδωσα διεξοδικές απαντήσεις. Θα σας στείλω στη συνέχεια πιο λεπτομεριακές απαντήσεις για ορισμένα θέματα που παρέλειψα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, στην Επίτροπο που ήρθε και αφιέρωσε χρόνο στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να μην είναι τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Προσβλέπουμε σε συνέχιση αυτής της συζήτησης και των επαφών. Ladies and gentlemen, may we continue? Uh, Παρακαλώ συνεχίζουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρώτο, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμανς, που είναι αρμόδιος επίτροπος, όπως ξέρετε, για την καλύτερη νομοθεσία, τις διοργανικές ε, σχέσεις, ε, το κράτος δικαίου και την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφάπτονται σε μεγάλο βαθμό οι αρμοδιότητε του με τι αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη νομοθεσία, την απλούστευση του ενωσιακού δικαίου, εφαρμογή και παρακολούθηση τη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και κυρίω επιλογή νομική βάση και σεβασμό τη αρχή τη επικουρικότητα και της αναλογικότητας, καθώς και ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για θέματα που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, δικονομικό δίκαιο και θέματα δικαστικής και διοικητικής συνεργασίας ε, σε αστικές υποθέσεις. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και η, πιθανή αναθεώρηση της Διοργανικής Συμφωνίας του 2003 για την ε, καλύτερη νομοθεσία. Άλλο θέμα που απασχολεί την Επιτροπή μας είναι εφαρμοστικές και καταξουσιοδότηση πράξης και συναφή νομικά προβλήματα. Μια και έχουμε μείνει ήδη πίσω στο χρόνο μας, θα δώσω χωρίς άλλη καθυστέρηση το λόγο στον πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια που έχουμε καθυστερήσει, προτείνω να περάσουμε απευθείας στις ερωτήσεις χωρίς να κάνω εγώ εισαγωγές. Now this is an original solution to the... Πρωτότυπη λύση στο πρόβλημα. Ο κύριος ε, Κωστόφ ε, ζητάει το λόγο από ό,τι βλέπω, ε. Mr. Kester, please. Äh, Κύριο Κάστορ, ευχαριστώ. Δύο θέματα θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα το ευρωπαϊκό ε, το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, το οποίο το συζητάμε εδώ και καιρό. Υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απογοητευτήκαμε γιατί μάθαμε πως έφυγε από την ημερήσια διάταξη της Κομισιόν και βεβαίως ε, ως ε, αρμόδιος ηγητής ε, σας απέστειλα και μία επιστολή. Σας παρακαλώ να το ξαναδείτε το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων να ξαναμπεί ε, επί Υπάρχουν κάποιες πτυχές που οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθούν όσον αφορά δηλαδή τον διαχωρισμό νομικής έδρας και μέρους όπου ασκούνται πραγματικά οι δραστηριότητες. Όχι, η έδρα πρέπει να βρίσκεται εκεί όπου ασκείται η κύρια δραστηριότητα. Και το άλλο θέμα είναι σε ποιο βαθμό η Κομισιόν θα μπορούσε να επανεξετάσει ε, το ζήτημα αυτό του δικαίου των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Το δεύτερον. Το τι γίνεται με τις διαιτητικές διαδικασίες στο πλαίσιο της ε, TTIP. Υπάρχει εδώ πρέπει μια γνωμοδότηση του Ζίγκφριντ Bros ο οποίος ήταν δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο και λέει πως θεωρεί πως η προστασία των επενδυτών, όπως λέγεται, αντιβαίνει και στο Γερμανικό Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τελικά παραβιάζει το σύστημα του διεθνούς δικαίου και εκτιμά πως μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, ΣΕΤΑ ή TTIP, με την ρήτρα αυτή για ακριβώς μια τέτοια διαιτητική διαδικασία δεν έχει καμία ελπίδα να σταθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πώς θα ήταν καλό λοιπόν να ζητήσουμε μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πριν συνάψουμε τέτοιες συμφωνίες. Ευχαριστώ κυρία Κάφμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο αφορά τις ε, εκτιμήσεις επιπτώσεων. Είπατε πως θέλετε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση εκεί πέρα. Θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς ε, τι σημαίνει αυτό και βεβαίως τι σημαίνει αυτό και κατά πώς θα μπορούμε να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία της Επιτροπής μας μετά. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό και σε μία ακρόαση και είπατε πως ε, το Κοινοβούλιο θα καταβάλει προσπάθειες ε, με τη δικιά του μελέτη επιπτώσεων αλλά δεν θέλει ούτε να τα ακούει το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω πως έχουν επαναληφθεί οι συζητήσεις και αν είχαμε καμία εξέλιξη ή κάτι άλλο το οποίο μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ε, για το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Είναι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο για να περάσει κάτι τέτοιο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ομοφωνία. Οπότε, ε, ε, αν έτσι έχει η κατάσταση, η Κομισιόν θέλει να είναι ρεαλιστική, να μην αφήσει κάτι τώρα να εκκρεμεί ε, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα να ληφθεί απόφαση στο Συμβουλίο. Εάν ήταν διαφορετικά τα μηνύματα ή αν χρειαζόταν ειδική πλειοψηφία, θα ήταν αλλιω Αλλά ε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πολλά κρατημέλη, όχι μόνο ένα, δεν θα συμφωνήσουν ποτέ με την πρόταση. Οπότε, ρεαλιστικά, η Κομισιόν αποφάσισε να το αποσύρει για το ISDS. Ε, ε, όπως τα λέτε, ε, ακούγοντας κανείς προσεκτικά, το παρουσιάζεται σαν κάτι το καινούριο τον ε, μηχανισμό αυτών διαιτησίας. Μα υπάρχουν δεκάδες, αν και περισσότερες διατάξεις σε εμπορικές συμφωνίες. Εάν ο νομικός αυτός που αναφέρατε έχει δίκαιο, τότε σε δεκάδες περιπτώσεις παραβιάζουμε το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ισχύει δηλαδή αυτό το οποίο λέτε. Του του Απέχουμε πολύ, οπωσδήποτε, από αυτό το οποίο θα θέλαμε ως μηχανισμό ISDS. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι σαφής. Δεν θα πω ναι σε ένα τέτοιο μηχανισμό, ο οποίος δεν θα λαμβάνει υπόψη τη θέση των Ευρωπαίων πολιτών του ε, πολιτισμού μας, του πώς έχουμε οργανώσει το νομικό μας σύστημα, την προστασία της πολιτιστικής μας ε, κληρονομιάς, ε, της παράδοσης, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο στις διαπραγματεύσεις μας. Και ξέρετε, εδώ ακριβώς πρέπει να είμαστε ισχυροί ως Ευρωπαίοι. Γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν παραδοσιακά πως ό,τι είναι καλό για τις είπα είναι καλό για τον κόσμο και αν γίνουν όλοι οι Αμερικάνοι θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Εντάξει, μπορεί αυτοί να το βλέπουν έτσι, αλλά διαφέρουμε. Έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες, αξίες ε, και πρέπει να γίνονται σεβαστά αυτά τα πράγματα και στην TTIP. Και αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά το να πούμε, περσέ, ότι ένα σύστημα τέτοιο όπως το ISDS είναι κατά των συνθήκων ή κάποιου συντάγματος είναι περίεργο δηλαδή αν δούμε πόσες διμερείς τέτοιες συμφωνίες έχουν τα κράτη-μέλη στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Για το θέμα των μελετών αντικτύπου. Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι πως κάνουμε αρχικά μελέτες αντικτύπου αλλά δεν κάνουμε όταν περάσει μια πρόταση και γίνει νομοθεσία. Και βεβαίως δεν αξιολογούμε τον αντίκτυπο του τελικού αποτελέσματος. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί ξέρετε καμιά φορά η Κομισιόν προτείνει ένα άλογο όπως λένε και προκύπτει καμήλα από την όλη διαδικασία μέσω Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και μπορεί τελικά η νομοθεσία να είναι τελείως διαφορετική από την αρχική πρόταση που αφορούσε η μελέτη αντικτύπου. Οπότε εγώ πάντα έλεγα, αν θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος, ε, πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του τελικού νομοθετήματος και για να γίνει αυτό ε, πρέπει ε, να εμπλακεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο κάτι κάνει. Έχει κάνει κάποια τέτοια βήματα το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Εγώ έχω υποβάλει αυτή τη θέση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω να τα λέω και στο Συμβούλιο και θεωρώ πως θα πρέπει να είναι επίσης αναπόσω στο τμήμα των διαπραγματεύσεων για τη Διοργανική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω πει επίσης πως το ιδεώδες είναι πως ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού τα τρία θεσμικά όργανα την αξιολόγηση αντικτύπου. Αν συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει μια λογική πράγματι να γίνεται μια αξιολόγηση που θα είναι ανεξάρτητη. Ε, ε, υπάρχει ένα συμβούλιο τέτοιο που θα είναι ανεξάρτητο από τα τρία αυτά ιδρύματα. Αλλά όσο δεν γίνεται αυτό, δεν βλέπω τον λόγο. Τούτου λεχθέντος οπωσδήποτε θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία με το να ορίσω εγώ ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πιο αξιόπιστοι ως προς ε, ακριβώς την ανεξαρτησία τους και από πολιτικές επιρροές. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Η πρώτη αφορά το πρόγραμμα εργασίας της ε, Κομισιόν. Ε, δεν καταφέραμε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα ήθελα να πω πως ε, η δικιά μας η ομάδα χάρηκε ιδιαίτερα όταν διάβασε το πρόγραμμά σας. Και έτσι να το πω και λίγο χήμα, ελπίζω να τα κάνετε αυτά τα οποία υπόσχεστε. Και τώρα λέτε πως απαιτείται μια ρεαλιστική προσέγγιση και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να πετύχουμε κάτι στο Συμβούλιο, τότε ας τα αφήσουμε κατά μέρος. Έχετε απολύτως δίκιο. Και θα ήθελα εδώ πέρα να σας υποστηρίξω πλήρως. Δεύτερο θέμα, καλύτερη νομοθεσία. Πράγματι πάρα πολύ βασικό για εμάς το Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ασχολούμαστε με εκθέσεις και ο συνάδελφος εδώ πέρα δίπλα μου. Εμείς πάντα ως Κοινοβούλιο ζητούσαμε να υπάρξει ένα ανεξάρτητο τέτοιο συμβούλιο σαν αυτό που ζήτησε και ο συνάδελφος και πάντα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση από Κομισιόν και Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν να σας παρακινήσω, να σας παρακαλέσω χρειάζεται ένα όργανο ανεξάρτητο το οποίο θα ελέγχει τις ε, προδιαγραφές και στην αρχή και στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας ε, να βλέπει λεπτομερώς ε, το αποτέλεσμα Γι' αυτό ακριβώς αναμένουμε από σας να μας πείτε τι άλλη άποψη έχετε. Και τέλος, στο πλαίσιο αυτό, τελευταία ερώτηση. Με μεγάλη χαρά διάβασα πως ο Έντμουντ Στόιμπερ, πρώην Πρωθυπουργός μου εκεί πέρα στη Βαβαρία, θα είναι ειδικό σας απεσταλμένος ε, θα έρθει και εδώ πέρα αύριο βεβαίως, θα τον ρωτήσω τι ακριβώς ε, θα κάνει, αλλά μπορείτε και να μας πείτε ποια θα είναι η αποστολή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γκούτλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τίμερμαντς, που ήρθατε. Το εκτιμούμε όλοι μας. Είναι χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις. Ξέρω ότι δεν χρειάζεται να σας πω την κατάσταση στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι 26 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι. 6 εκατομμύρια από αυτούς είναι νέοι. Και 125 εκατομμύρια ζουν κάτω από τον κίνδυνο της ε, φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχουν ανισότητες, ε, υπάρχουν προβλήματα κοινωνικού dumping και προβληματικές συνθήκες εργασίας, ασταθής εργασία. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ευρώπη. Είναι μια ορολογιακή βόμβα αυτή, η οποία οξύνει τους κινδύνους ε, πολιτικών ε, διεκδικήσεων ακραίων στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ό,τι κάνει η Κομισιόν και ό,τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιδράσει. Πιστεύω ότι έχετε μια καλή ατζέντα. Φοβάμαι λιγάκι όμως ότι η Κομισιόν δεν ξέρω πώς θα εξισορροπήσει τις, α, τις πολιτικές δυνάμεις ό,τι αφορά την νομοθεσία που θα προωθήσει. Ε, θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθος. Δίδεται μεγάλη προσοχή σε αυτό. Καλή είναι η πρόθεση, αλλά μην ξεχνάτε τον κίνδυνο ο, του να περάσει νομοθεσία πολύ λεπτομερής, πολύ τεχνική. Ο κόσμος και τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι είναι υπερβολικά τεχνική νομοθεσία. Επίσης φοβάμαι ότι αν προσπαθήσουμε πολύ να μειώσουμε το κόστος παρά να πετύχουμε κάποιους στόχους, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές ανισότητες, Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην πράσινη ατζέντα. Η ισορροπία είναι πολύ λεπτή. Ποια είναι η πρόθεσή σας, πώς θα εξισορροπήσετε όλα αυτά τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, ούτως ώστε η μείωση της γραφειοκρατίας να μην υποσκάψει τη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την περιβαλλοντική προστασία, την ε, ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ. Ευχαριστώ κύριο Ντεγκράντες. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Θεωρήστε ο εγκέφαλος της Επιτροπής ιούνκερ Από τις αρχικές ερωτήσεις που θέσαν όλοι σε σχέση με το έθνομοθετήν, ε, και την προσπάθεια που κάνετε προς αυτήν την κατεύθυνση, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ. Αλλά πρέπει να σεβαστείτε την επικουρικότητα. Είναι μια αρχή που μας έχει εμπνεύσει. Να νομοθετούμε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, πιο κοντά στον πολίτη. Συμφωνώ με όλα αυτά. Τέλεια είναι. Δεν θεωρείτε, κύριε Τίμερμανς, ας πούμε, τι έγινε στην προηγούμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Ε, όταν έχουμε λιγότερη νομοθετική εργασία, θα ελέγξουμε περισσότερο την εκτελεστική εξουσία. Αλλά υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Ένας αναπότρεπτος πειρασμός. Μπορεί μέσω της Κομισιό να ασκηθεί έλεγχος στις κυβερνήσεις για το έργο τους. Εσείς ε, ξέρετε τι πρέπει να γίνει ως νομικός βέβαια. Η ερώτησή μου μετά από όλα αυτά είναι η εξή. Θα θυμάστε αυτές τις απόπειρες στο Παρίσι. Και όλοι μας διαπιστώσαμε κάτι που εμείς ξέραμε στην Ισπανία, γιατί είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτό, ότι η τρομοκρατία έχει παγκόσμια εμβέλεια. Ε, συνδέεται με τη μετανάστευση με τη Συμφωνία Σέγγεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση της ε, ελευθερίας αλλά και μια άλλης αξίας που είναι η ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει στην κορυφή όλης της προσπάθειας αυτής να θέσουμε τους πολίτες. Αυτό σημαίνει εξασφάλιση της ασφάλειάς τους. δεν θα πρέπει να ξαναδούμε τις προτεραιότητές μας ή εν πάση περιπτώσει να δούμε τι θα κάνουμε το θέμα της μετανάστευσης και της διατήρησης των ελευθεριών και της ασφάλειας και της, το πώς αντιμετωπίζουμε την παγκοσμιοποιημένη τάση που δείχνει σήμερα η τρομοκρατία. Την παγκόσμια διάσταση, αν θέλετε, της τρομοκρατίας. Um, Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά το εφνομοθετήν, τη βελτίωση της νομοθεσίας ε, σε συνδυασμό με το έργο του κυρίου Στόιμπερ. Ένα θέμα συναφές με αυτό που είπατε και εσείς. Πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία χωρίς ε, να υπονομεύσουμε άλλους στόχους που έχουμε. Γιατί όσοι λένε ότι θέλουν να μειώσουμε τη, ε, τη γραφειοκρατία, δεν θέλουν να μειώσουμε και την κοινωνική προστασία, την περιβαλλοντική προστασία αλλά έτσι μερικές φορές έχει διατυπωθεί και από την αρχή όταν άρχισα να μιλώ για γραφειοκρατία και στη δική μου πολιτική οικογένεια λένε «Α, θέλετε να υπονομεύσετε την περιβαλλοντική προστασία και να φημώσετε ή να καταργήσετε την κοινωτική προστασία. Σε καμία περίπτωση δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο και αυτό είναι το ζητούμενο. Και στα τελευταία χρόνια αν δείτε τι έγινε με την ευρωπαϊκή ολοκληρωσή, από πού έχουμε την ισχυρότερη στήριξη, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιλήφθηκαν ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πού χάσαμε την τελευταία πενταετία κάθε υποστήριξη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάλι και στόχος μου είναι να ξανακερδίσω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για την Ευρώπη και υπέρ της ολοκλήρωσης. Γιατί αν μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κάνουν περισσότερες προσλήψεις. Αν μειώσουμε τις ε, γραφειοκρατικές διατυπώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερο χρόνο ε, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι στην ε, συμπλήρωση εγγράφων και διοικητικών διατυπώσεων. Και έτσι θα αυξηθούν οι προσλήψεις, θα αυξηθούν ε, οι θέσεις απασχόλησης και άρα η αξιοπρέπεια. Και θα πρέπει αυτά τα 26 εκατομμύρια να μπορεί να κάνει τις επιλογές του και να ανακτήσει την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Είναι σκανδαλώδες που σε μερικές χώρες μέλη πάνω από το μισό του πληθυσμού κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι και αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι από την κοινωνία. Είναι φρικτό που τόσοι άνθρωποι δεν μπορούν πια να μείνουν μόνοι τους και να συντηρηθούν και επιστρέφουν στην οικογενειακή αιστεία, στο πατρικό του σπίτι. Και έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση από το 1930, που έχει μετατραπεί σε κοινωνική κρίση σε πολλές χώρες μέλη και τροφοδοτεί τα ακραία και εξτρεμιστικά κόμματα και ξεσηκώνει τους ανθρώπους και αρχίζει και αναβιώνει τους παλιούς ευρωπαϊκούς δαίμονες ε, και την επίρρηψη ευθυνών σε άλλους. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τους αποδιοπομπαίους τράγους. Ε, στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό και η μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση των θέσεων απασχόληση είναι ένας τρόπος καταπολέμησης του εξτρεμισμού. Φαίνεται τεχνικό θέμα, αλλά πραγματικά είναι συνυφασμένο με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών μας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λέει ότι το σχέδιο Juncker μπορεί να λειτουργήσει και μάλιστα να αξιοποιηθεί και να... Αλλά πιστεύει ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα ενισχυθεί με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Το λέει ίδια η Τράπεζα Επενδύσεων και την πιστεύω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη μείωση των κοινωνικών ή των περιβαλλοντικών μας στόχων. Σε καμία περίπτωση το ένα δεν συνεπιφέρει και το άλλο. Πάντως το Συμβούλιο δεν θα καταλήξει συμφωνία για ένα ενιαίο έντυπο ΦΠΑ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχει κανείς μια μικρομεσαία επιχείρηση και έχει εμπορικές συναλλαγές με 3-4 κράτη-μέλη και κάθε φορά πρέπει να συμπληρώνει διαφορετικά έντυπα, αυτό είναι γραφειοκρατικό άχθος, διοικητικό άχθος που θα μπορούσαμε να το καταργήσουμε αν ήμασταν σοβαροί στο στόχο μας. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βοηθήστε με για να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν απίστευτο όταν άκουσα ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει καν για ένα ενιαίο έντυπο πανευρωπαϊκό για το ΦΠΑ. Ούτε καν γι' αυτό. Πάντως ε, θα συνεργαστούμε με τον κύριο Στάιμπερ για τα θέματα αυτά. Τώρα, θέμα επικουρικότητα και νέων προτεραιοτήτων. Ένας πρώην ε, Βρετανό Πρωθυπουργό, όταν ερωτήθηκε για τι προτεραιότητε του, είπε ο Μακμίλαν, τα γεγονότα αγαπητέ τα γεγονότα. Μπορεί κανεί ε, να εκπονεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ναι, αν έχουμε ένα εξωτερικό γεγονό και κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση, μια απειλή, θα πρέπει να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων και να βρούμε λύσει ε, και να δώσουμε απαντήσει στι απειλέ που ε, είδαμε στο Παρίσι, που ουσιαστικά απειλούν τον ιστό τη κοινωνία. Δεν είναι μια απλώς τυχαία τρομοκρατική επίθεση ενέργεια. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια επίθεσης κατά των θεμελιωδών αξιών που εστερνιζόμαστε εμεί οι Ευρωπαίοι. Και θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την απειλή και μάλιστα κατά προτεραιότητα. Είναι υποχρέωσή μας. Κανένας δεν θα πει συγγνώμη, δεν είναι στι προτεραιότητές μας, ελάτε του χρόνου. Προφανώ και όχι. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν μαζί σα ότι αν κάτι θα πρέπει να κάνουμε, πρέπει σίγουρα να ανταποκριθούμε και θα έχουμε και ένα άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Φεβρουάριο με αυτό το θέμα. Γιατί όλοι είμαστε οι συνυπεύθυνοι και φυσικά πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να υπησέλθω σε συζήτηση με τα κράτη-μέλη για αρμοδιότητες στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν θα πρέπει να φαγωθούμε μεταξύ μας. Οι πολίτες θέλουν λύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη-μέλη όπως μπορεί και με κάθε τρόπο στα πλαίσια της εντολής και της αρμοδιότητάς της για να δώσουμε μια επιτυχημένη απάντηση και σωστή απάντηση σε αυτές τις απειλές. Και ένα ακόμη σχόλιο. Ο μόνος τρόπος που θα λειτουργήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και το σεβασμό όλων των χωρών μελών για το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είναι ο πυρήνας ευρωπαϊκής συνεργασίας. Φυσικά χρειαζόμαστε επεγνωσμένα την ελευθερία έκφρασης. Αν καταργήσουμε την ελευθερία έκφρασης παλιδρομούμε στην κατάσταση πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό θα είναι το τελευταίο που θα χρειαζόμασταν 70 χρόνια μάλιστα μετά το Auschwitz. Και αν δεν θέλουμε να επαναληφθεί το παρελθόν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε κάθε μειονότητα να αισθάνεται ασφαλής ε, και προστατευμένη στην Ευρώπη. Αυτό με κρατάει εξάγρυπνο αυτή τη στιγμή. Το γεγονό ότι και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο η πλειοψηφία της ευρωπαϊκής κοινότητας ε, έχει κάνει ανάλυση και είπε ότι δεν βλέπει μέλλον για αυτήν στην Ευρώπη. Και αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο, μπορούμε να μιλάμε μήνες και χρόνια για καλύτερη νομοθεσία, αλλά θα υποστούμε πολλά δεινά από κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Φυσικά και υπάρχουν και νέες προτεραιότητες με βάση τις νέες εξελίξεις και θα τα αποκριθούμε και σε αυτές. Και σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταθεί στο ύψος των προκλήσεων. Θα ήθελα να σας πω από την αρχή να, για να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, να μην κάνουμε καν ερωτήσεις, αλλά να πείτε τις απαντήσεις. Από τη στιγμή που διοριστήκατε, ε, σας εκτιμούν πάρα πολλοί προβουλευτές για το, τη σοβαρότητα με την οποία κάνετε αυτό το διάλογο. Άκουσα αυτά που είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από λίγες ε, μέρες σας έδωσα την ευκαιρία να μας δώσετε λεπτομέρειες για τα τρία πράγματα που θα κάνετε μέσα σε 12 μήνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο είπατε και τεκμηριώσατε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και παραπάνω, και κάτι παραπάνω από αυτό. Θέλω να σας ξαναδώσω λοιπόν την ίδια ευκαιρία και ελπίζω να την αδράξετε. Τώρα, δεύτερον, σε σχέση με το, την ατζέντα που έχουμε για την έξυπνη νομοθεσία. Εγώ ήμουν εισηγητή στην Επιτροπή αυτή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερω που θεωρείται ότι πολύ από το έργο που κάναμε εμείς ε, είναι άξιο για να ενσωματωθεί στο δικό σας ε, έργο ε, και είναι σημαντικό αυτό για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στο μέλλον. Και πολύ επικοδομητικά είπατε ότι αν χρειαστεί, οι υπάλληλοι τη Κομισιόν θα πάνε στα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτω ώστε να του δώσουν περαιτέρω ε, εξηγήσει και οδηγίε για το πώ θα προχωρήσουν. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή σε αυτό. Για να χρησιμοποιήσω τα δικά σα λόγια. Συχνά συμβαίνει, πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, να στέλνουμε ένα άλογο στα Εθνικά Κοινοβούλια. Μερικά δεν το δέχονται και μερικά παρουσιάζουν του πολίτε του, το παρουσιάζουν ω καμήλα και λένε εμεί το στείλαμε. Ε, μερικές φορές ε, ε ενσωματώνται διαφορετικά ή μάλλον ε, εφαρμόζεται διαφορετικά η, ευρωπαϊκή νομοθεσία ή παρουσιάζεται διαφορετικά στους πολίτες κτλ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Το θέμα του αλόγου και της καμήλας ε, αφορούσε κάτι άλλο, γιατί ξεκινάει κάτι ως άλογο και μετά από επεξεργασία στο Συμβούλιο και στο κοινοβούλιο μετατρέπεται σε καμήλα. Αυτό που είπατε, το πώς παρουσιάζουν μερικές φορές τα κοινοβούλια στην κοινή γνώμη το θέμα είναι κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα τώρα κύριε Αντιπρόεδρε να σας κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ας ε, κάνουμε μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αν κατάλαβα καλά, το ιδανικό για σας θα ήταν ε, κοινή, ανεξάρτητη αξιολόγηση, αντικειμενική, που θα γίνεται από εμπειρογνώμονες ε, τελείως ανεξάρτητους από μας. Για να γίνει η μελέτη των επιπτώσεων και των ε, αποτελεσμάτων εγγραφών, εγγράφων συγγνώμη, που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Γιατί αυτά ε, τα έγγραφα στη συνέχεια θα εγκριθούν και θα αποτελέσουν τον κορμό του ενωσιακού δικαίου. Αυτό όμως δεν είναι δυνατό χωρίς ε, συμφωνία του Συμβουλίου. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να πάμε ακόμη πιο μακριά και να πούμε ότι αν έχει το Κοινοβούλιο πρόβλημα, με δική μας ε, έγκριση να κάνουμε αυτή τη μελέτη του αντικτύπου, αυτή τη μελέτη των αποτελεσμάτων. Για να δούμε δηλαδή ε, πώς θα εξετάσουμε αυτό το ζώο και τι μορφή θα λάβει τελικά όταν έχει ξεκινήσει από μία μορφή και μετατρέπεται σε άλλη στην πορεία. Επίσης, άλλο σημαντικό θέμα είναι η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και η ενσωμάτωσή του στην ε, εσωτερική τάξη, την εθνική τάξη. Εκεί έχουμε προβλήματα με την τήρηση των προθεσμιών για την ε, εμπρόθεσμη εφαρμογή, για τη σωστή εφαρμογή, για τη βούληση εφαρμογής μερικές φορές. Και μπορεί μια χώρα να δέχεται καταρχήν μια νομοθετική ρύθμιση, αλλά μετά να μην εφαρμόζεται στην εσωτερική εθνική νομοθεσία. Είναι πραγματικά σαν να προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο μερικέ φορέ. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποιους μηχανισμούς ώστε να μπορέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου εθνικά. Επίσης γνωρίζετε από όλοι εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την βλέπουμε εμείς, διαφέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπουν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται περισσότερο για την ελεύθερη υλοποίηση των στόχων της ζωής τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Χάρτα θεμελιώδη Δικαιωμάτων και με βάση κάποιες άλλες διατάξεις που θα είναι καλές και θα εφαρμόζονται σωστά. Μερικές φορές όμως οι συμπολίτε μας δημιουργούν κακή γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της εντύπωσης που δίνεται από κάποιους πολιτικούς και από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εχθρικά προς την Ένωση και επικεντρώνονται σε κάποια νομοθετικά παράδοξα που είτε έγιναν είτε προ προβλέπουν ότι θα γίνουν στο μέλλον. Οπότε, ε, θα πρέπει σωστά να εκπονήσουμε το κοινοτικό δίκαιο, τι θα γίνει στο μέλλον και επίσης ε, να γίνει μια υποπτία και μια επισκόπηση της ε, ισχύω της νομοθεσίας και το κατά πόσο εφαρμόζεται στις εθνικές ένωμες τάξεις. Γιατί εκεί έχουμε μερικές φορές μερικά παράδοξα και αστεία φαινόμενα. Εκεί θα πρέπει να βρούμε κάποια λάθη και να τα διορθώσουμε. Ε, και χαίρομαι που δώσατε χρόνο για περισσότερη συζήτηση γιατί έχουμε περισσότερα νομοθετικά σχέδια και προτάσεις. Καλό αυτό για την αρχή, αλλά αυτό θα είναι το κλίμα που θα επικρατήσει όλη την πενταετία. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχω δύο ερωτήσεις ε, για εσάς. Η πρώτη αφορά τον Ευρωπαϊκό Δικονομικό Κώδικα. Το 2013 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν μία πρόταση κανονισμού για το δικονομικό διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα καθόριζε τις γενικές αρχές που ρυθμίζουν τις ε, δραστηριότητες ε, των θεσμικών οργάνων. Τότε η Κομισιόν απάντησε πως είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μελετούσε προσεκτικά πριν αναλάβει ε, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στο μέτωπο του ε, οικονομικού δικαίου. Κατόπιν Κύριε Τίμερμανς, οπωσδήποτε θα ξέρετε το εντατικό lobbying που λαμβάνει η χώρα και στο οποίο ασκείται κριτική κυρίως ε, λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Ταυτόχρονα οι επαφές μεταξύ θεσμικών οργάνων, ΜΚΟ και επαγγελματικών οργανώσεων και κλαδικών οργανώσεων συνεχίζονται γιατί έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη ορθών πολιτικών πολιτικών σωστών για τη δημοκρατία και την ενιαία αγορά. Το δεύτερο μου ερώτημα λοιπόν αφορά την διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό μητρό διαφάνειας, το οποίο είναι στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2015 και έχει πράγματι ε, φτάσει η ώρα να μου πω ότι έχουμε αργήσει κιόλας. Ε, το ερώτημα μου είναι λοιπόν πότε θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και με ρωτήσατε για τις τρεις προτεραιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φοβάμαι πως ε, θα σας δώσω την ίδια απάντηση και πάλι. Πρώτον, οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μας έδωσαν 10 πράγματα που τους ενοχλούν. Και θέλουμε η Κομισιόν να αναλύσει αυτό τον κατάλογο και να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν διαλέξω εγώ τρία πράγματα, από τα δέκα θα είναι μάλλον λάθος. Δεσμεύομαι όμως πως θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να προσπαθήσω να τις βοηθήσω με όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά τα 10 σημεία αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος ε, να δούμε τι είναι εφικτό. Αλλά το μελετάμε. Ε, και σας διαβεβαιώ πως έχει την αμέριστη προσοχή μου το θέμα αυτό, γιατί όπως σας είπα θεωρώ πως πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να δημιουργήσει θέσεις εργασίας έτσι ώστε ο φούρναρης ε, και ο οικοδόμος και ο εργολάβος οικοδομών να θεωρούν πως ε, δρούμε προς το συμφέρον τους. Ένα πρόβλημα βεβαίω που είναι κοινό για όλους εμάς πολιτικούς ε, και το είδα αυτό στην ΚΟΖΑΚ είναι πως ε, συνέχεια πολιτική ασχολούμαστε για, με το μέλλον και το τι θέμα να κάνουμε στο μέλλον και όλα αυτά αλλά ποτέ δεν ασχολούμαστε με το τι ακριβώς ε, θεωρούμε, τι, με το τι ακριβώς χρειάζονται οι πολίτες και θα είναι οι πολίτες. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ο καθένας γράφει ό,τι θέλει όταν μεταφέρονται οι οδηγίες στην εθνική νομοθεσία. Έχει φτάσει νομίζω η ώρα να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη με τη δική σας τη βοήθεια να κοιτάξουν το τι υπάρχει ήδη στα κράτη-μέλη και να δουν πώς χρειάζεται να καταργηθεί κάτι, να αλλάξει κάτι, να απλοποιηθεί κάτι άλλο. Νομίζω πως η αχίλιος πτέρνα της πολιτικής είναι πως ε, δεν είναι το δυνατό μας σημείο η λογοδοσία για τα όσα κάναμε στο παρελθόν θα έλεγα. Και έχει φτάσει πια η ώρα η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία να επανεξεταστεί. Νομίζω πως έχουμε ένα καλό παράδειγμα τώρα που δίνει η Επίτροπος Γεωργίας. Και νομίζω πως εάν μιλήσουμε με τα κράτη-μέλη θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Επίσης, οι επιπρόσθετες διατάξεις είναι σοβαρό πρόβλημα. Κάποια κρατημέλη κάτι κάνουν, κάποια άλλα όχι. Ελπίζω πως στενή συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών ε, κοινοβουλίων ε, να καταλήξουμε σε κάποιους τρόπους για να καταπολεμήσουμε αυτή την πρακτική. Και αντιλαμβάνομαι πως ε, υπάρχει και στην ΚΟΣΑΚ μια προσπάθεια να δημιουργηθεί με πλατφόρμα για αυτό το λόγο. Τώρα για το Συμβούλιο Αξιολόγησης Αντικτύπου να είμαι σαφής. Σε αυτή τη φάση το βάρος είναι στην Κομισιόν για την πρόταση που θα καταθέσει. Ε, οπωσδήποτε παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτή την ευθύνη. 40% των προτάσεων επιστρέφεται γιατί ε, όπως ξέρετε η αξιολόγηση αντικτύπου είναι ευθύνη των υπηρεσιών και όπως σας είπα 4 στις 10 περιπτώσεις επιστρέφονται ως απαράδεκτες γιατί δεν είναι ικανοποιημένο το Συμβούλιο αυτό. Θα ενισχύσω την ανεξαρτησία στη στελέχωση του Συμβουλίου αλλά πρέπει να παραμείνει θεωρώ εντός της Κομισιόν μέχρι να φτάσουμε σε μια δυνητική κατάσταση στο μέλλον όπου θα συμφωνήσουν και τα τρία θεσμικά όργανα για την εξέταση και του τελικού προϊόντος μετά την νομοθετική διαδικασία γιατί τότε μπορούμε να αξιολογήσουμε το ποιος είναι ο αντίκτυπος των ε, κρατών μελών. Αυτά τώρα δεν σας λέω τίποτα το καινούριο αλλά νομίζω καλό είναι να το πούμε Κάποιες φορές ε, στις διαπραγματεύσεις μας, ε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, η επιθυμία για συμβιβασμό είναι ισχυρότερη από το να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι περιττό βάρος με αυτό το συμβιβασμό. Δεν το αμφισβητεί νομίζω κανείς. Και νομίζω πως ε, αν γίνεται μια αξιολόγηση αντικτύπου στο τέλος θα πούμε το εξής ναι εντάξει βρήκαμε ένα συμβιβασμό αλλά κοιτάξαμε το τι σημαίνει όσον αφορά το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα στο κράτος μέλος και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου αν το κάναμε αυτό θα ε, ξανακοιτάζαμε τις συμβιβαστικές λύσεις που βρήκαμε. Τώρα, συμφωνώ πως η εικόνα που υπάρχει για την Ευρώπη στη δημόσια συζήτηση είναι συχνά άδικη. Δεν αξίζει αυτή η εικόνα στην Ευρώπη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η εικόνα και άδικη να είναι υπάρχει και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να την τροφοδοτούμε και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε κάποια ρεαλιστική εικόνα για να διορθώσουμε την αδική εικόνα. Παραδείγματο χάρη. Ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούστηκε για τον οικολογικό σχεδιασμό, το οποίο ε, το γελιοποιούν ε, συχνά, ξέρετε, μέχρι την ίσα ε, απαγωγή. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει και ο Βρετανικός τύπος που λέει πως ε, είναι γελίο το ότι η Ευρώπη λέει πως πρέπει να σβήνουν οι συσκευές αυτομάτως μετά από μισή ώρα και μετά στο τέλος του άρθρου λένε εντάξει δεν είναι και τόσο γελίο, γλιτώνει ενέργεια, λεφτά κτλ. Οπότε, Εάν υπάρχει ευκαιρία να αναπτύξει κανείς τη λογική του, θα δημιουργηθεί μια διαφορετική εικόνα. Δεν έχω ακόμα απελπιστεί εντελώς. Μετά. Μιλήσατε για την έκθεση Berlinguer και το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο. Το είπα στην ακρόαση και αυτό ισχύει και για την ε, Κρυσταλίνα Γεωργιέβα πως η Κομισιόν οπωσδήποτε θα το εξετάσει αυτό. Το τι θα γίνει τώρα αυτό, σε τι στόχο θα μεταφραστεί για το διοικητικό δίκαιο δεν το ξέρω. Για το lobbying τώρα. Εγώ θα χαιρόμουν αν το Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη, αποφάσισε να έχει πλήρη διαφάνεια στο ποιους συναντούν οι βουλευτές και αποφάσιζαν να συναντάνε μόνο άτομα τα οποία είναι σε ένα μητρό, όπως ισχύει για τους επιτρόπους και τα μέλη του ιδιαίτερου γραφείου τους χρειάζεται η διαφάνεια νομίζω και στα θεσμικά όργανα και είναι η προστασία μας ε, από παρερμηνία της δουλειάς μας και πιστεύω πως ε, δεν μπορεί ε, να γίνεται κάτι εντός της Κομισιόν του Κοινοβουλίου χωρίς να ενημερωνόμαστε όλοι από τους ενδιαφερόμενους. Αλλά η εντύπωση πως υποκύπτουμε σε αυτούς την αποκαταπολεμάται μόνο με την πλήρη διαφάνεια. και θα το προωθήσω αυτό και ελπίζω η Επιτροπή σας να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας ε, για να προηγηθεί το Κοινοβούλιο και να ακολουθήσει το Συμβούλιο. Okay. Uh, five minutes. Uh, I'm, running out of time because I'm... Δεν έχω αρκετό χρόνο σε 20 λεπτά πρέπει να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της ε, Ιαπωνίας. Θα πρέπει να πάω πίσω στο γραφείο μου στην Κομισιόν. Αν θα μπορούσα να κλείσω εδώ τη συζήτηση σε 5 λεπτά θα με βοηθούσατε πολύ. Να επιτρέψουμε δύο ακόμα ερωτήσει. Κυρία Χαουτέλα. Χαουτάλα. Άκουσα αυτά που είπατε για την έκθεση Berlinguer και τις συνέπειες. Ε, ήμουνα εισηγήτρια ε, για αυτό το θέμα και χαίρομαι για την ανοιχτή σας τάση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει αυτό να φέρει προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα όσα έχουμε τώρα δηλαδή. Συμφωνώ επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα ήταν πολύ πιο πιστικό αν ξεκινούσε από τη δική του τη διοίκηση αυτές τις αλλαγές. Έχουμε τη δυνατότητα. Ε, περιμένω να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες σας γι' αυτό και ελπίζω να βρούμε έναν δρόμο προς τα εμπρός. Θα ήθελα ακόμα να κάνω μια ερώτηση. Πήγα Διάβασα το εγγράφο της Κομισιόν για το TTIP και εντυπωσιάστηκα από τη γενική έκθεση που προέκυψε από τον 7ο γύρο διαπραγματεύσεων. Δεν θα πρόκειται να μιλήσω εδώ πέρα για τα μυστικά, αλλά υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις για το διοικητικό δίκαιο και τις διαφορές μας. Τώρα που θα κάνουμε και μια ακρόαση όπου θα συγκρίνουμε το διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, την ακρόαση αυτή θα την κάνουμε σε λίγες εβδομάδες, καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε λίγα για αυτές τις διαφορές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, στην ακρόασή σας μας είχατε πει ότι θα είσαστε παρόν εδώ στο Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, γιατί όπως ε, και στον έρωτα ε, πρέπει να δίνουμε αποδείξεις αυτού του, πράγμα, του πράγματος. Στην Αργεντινή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να διαλέγει τα πουρα του και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να γυαλίζει τις μπότες του δεν είναι κακός άνθρωπος. μετά τα 90 κείμενα που μπλοκάρατε, πιστεύετε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια εξέβρεσης ανάπτυξης, τη οδού για την ανάπτυξη. Έχετε τη δυνατότητα για την, για την ιδέα αυτού του δημοσιονομικού φιδιού, ε, όπως είχαμε κάνει ε, με την ε, Επιτροπή Βέρνερ το 1975, είχαμε βάλει αυτό το φίδι για να μειώσουμε τις διαφορές που υπήρχαν, δημιουργούσαν πρόβλημα στην οικονομία. Τώρα, για την ε, καυτή επικαιρότητα που αναφέρατε προηγουμένω, ε, μιλώντα με μερικού ε, συναδέλφου, η απόπειρα στο Παρίσι δεν είναι μόνο θέμα τη Γαλλία. Υπήρχε το 2004 η Μαδρίτη και το Λονδίνο το 2005. Νομίζω ότι ήγηκε η ώρα δυστυχώ για να δημιουργηθεί μια καλύτερη οργάνωση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Έχετε την ε, πρόθεση να επεξεργαστείτε νέες ιδέες ούτως ώστε να πιάνουμε τους ενόχους και να τους ε, διώκουμε και να τους δικάσουμε πιο αποτελεσματικά. Για τη διαθεσμική συμφωνία, για το εφνομοθετή, θα μας, μπορούσατε να μας πείτε το χρονοδιάγραμμα, γιατί θα θέλαμε εμείς ως Επιτροπή να ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή αμέσως. Για το διοικητικό δίκαιο. Δεν το ξέρω καλά το θέμα. Δεν το ξέρω καλά το θέμα του διοικητικού δικαίου. Δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία πληροφοριών, τις ε, νομοθετικές διαδικασίε, τέτοιου τύπου πράγματα μεταξύ και Αμερικανών. Είναι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα που διαπραγματευόμαστε με του Αμερικανού, βλέπουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε σε πολλού τομεί σε ό,τι αφορά το κανονιστικό μα πλαίσιο. Οποιαδήποτε συμφωνία με του Αμερικανού θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτέ τι ε, διαφορέ. Και δεν μπορούμε να τι επιλύσουμε. Θα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο όπου θα σεβόμαστε αμοιβαία τις διαφορές του ένας του άλλου. Και τώρα που μπαίνουμε στην καρδιά του θέματος, στο ψητό, βλέπουμε πόσες δυσκολίες υπάρχουν, αλλά αυτό είναι απαραίτητο. Εάν κάνουμε ό,τι πρέπει, νομίζω αυτό θα είναι σημαντικό και για τον υπόλοιπο κόσμο. Θα είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν κάποιοι να παντρέψουν διαφορετικά συστήματα χωρίς εμβιβασμούς, Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Αλλά είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το αν θα ξαναδούμε τις προτεραιότητες και την νομοθεσία μας, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Ε, αυτό είναι το τμήμα του προγράμματος REFIT. Και όπως είπα την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, ελπίζω να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάποια στιγμή την Άνοιξη τις ιδέες μας για το τι θα πρέπει να είναι σε αυτό το πρόγραμμα REFIT. Και σχέδια νομοθετη... νομοθετημάτων, αλλά και πώς μπορούμε να θεωρήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πιέρ Μοσκοβισή ε, εργάζεται πολύ έντονα για μέτρα για να αποφύγουμε το φορολογικό dumping, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι θα κάνουμε πρωτοβουλίες φέτος και ο Μοσκοβισή ασχολείται με αυτό το θέμα. Τώρα, τι μορφή θα πάρει αυτή η προσπάθεια, δεν ξέρω, είναι τα χωράφια του Πιέρ Μοσκοβισή, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούμαστε. Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, όπως σας είπα, επαναλαμβάνω ότι η Κομισιόν είναι στην υπηρεσία των κρατών μελών, θέλει να τα βοηθήσει να συντονιστούν καλύτερα, να εργαστούν μαζί καλύτερα. Καλό θα ήταν για την Ευρώπη αν προωθούσαμε την πρωτοβουλία να εξευρωπαίσουμε τη δικαιοσύνη, αν θέλετε. Και να λέμε ότι η Κομισιόν θα έχει την ε, ευθύνη. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε την ευθύνη, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τι συνθήκε, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη συνεργασία με τον Ευρωπα... μεταξύ των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων, ούτω ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη. Ε, το, σύστημα, το δικαστικό σύστημα μια χώρα, η ένωμη τάξη μια χώρα, θα πρέπει να σέβεται την ένωμη τάξη μια άλλη χώρα. Και με τι ιδέε μα θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Το πιο δύσκολο ερώτημα που άκουσα σήμερα ήταν αυτό του Προέδρου. Θέλει να του δώσω ημερομηνίε για το για το πότε θα έχουμε διαθεσμική συμφωνία για το εθνομοθετή. Και εγώ βιάζομαι, αλλά δεν νομίζω ότι βιάζεται το Συμβούλιο και δυστυχώ το χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστώ με το Συμβούλιο για να το πίσω να αρχίσει να κουνιέται. Η Λετωνική Προεδρία ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε καλά και όσο πιο γρήγορα μπορώ θα επανέλθω με μία απάντηση. Βασιστείτε πάνω μου. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Κάποια στιγμή θα επανέλθω και θα τα ξαναπούμε. Κύριε πρώτε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε που προλάβατε και ξεκινήσαμε αυτό το ζωντανό διάλογο. Ελπίζω κάποια στιγμή σύντομα να τα ξαναπούμε, γιατί βλέπετε πόσο ζωηρό είναι το ενδιαφέρον. Ladies and gentlemen, may... Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, θα συνεχίσουμε με το σημείο 7 της της διάταξης. και να καλωσορίσω θερμά την κυρία Νταϊάννα Γόλης, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, πρώην ε, Ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα με μια ηρωική προσπάθεια κατάφερε να έρθει παρόλα αυτά συνεδρίαση παρά τα προβλήματα της Eurostar. Ήρθε λοιπόν από το Λονδίνο και τη συνοδεύουν ο καθηγητή Βέντερχορστ, που είναι αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, του ELI και ο κύριο Χεφ Βαν Ερπ, που είναι μέλο τη εκτελεστική επιτροπή του ELI, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου. Πριν δώσω το λόγο στην Ταϊάννα Γόλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο που με προσκάλεσε στην ε, Γενική Συνέλευση που έγινε το περασμένο Σεπτέμβριο στο Ζάγκρεπ. Και μάλιστα είχαμε και στο εστιατόριο Γκράς Καβάνα ένα καταπληκτικό δείπνο. Μου έμεινε αξέχαστο. Ο λόγος λοιπόν στην πρόεδρο του ΙΕΛΑΙ, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, την κυρία Νταϊάννα Γόλης. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Είναι ευχαριστησή μου που βρίσκομαι εδώ ξανά με διαφορετικό ρόλο. Είναι βεβαίως τιμή μου, χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και με τους συναδέλφους, τους δύο καθηγητές. Αντιλαμβάνομαι πόσο χρόνος πιέζει. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να μοιραστώ μαζί σας και με τους συναδέλφους κάποιες σκέψεις για το τι είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου και το πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε ίσως με κάποια από τα προβλήματα που ανέφεραν και οι δύο επίτροποι. Πρώτα απ' όλα, τι είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου. Είναι ένα νέο θεσμικό όργανο τεσσάρων ετών που βασίζεται στο αντίστοιχο Αμερικανικό Ίδρυμα που υπάρχει εδώ και 100 χρόνια και βοηθάει το νομοθετικό έργο στις ΗΠΑ. Ποιοι είμαστε, είμαστε κάποιοι δικηγόροι, ο Χαμάν. Αλλά, να είμαι σαφής, δεν είμαστε κάποια οργάνωση ή λόμπι δικηγόρων, κάθε άλλο. Είμαστε ένας οργανισμός δημοκρατικός ε, διαφόρων δικηγόρων, μαχόμενων δικηγόρων, ε, δικαστικών επιμελητών, ε, καθηγητών πανεπιστημίου, όλη η νομική κοινότητα με μέλη από την Ευρώπη και παραπέρα. Και δεν έχουμε στόχο μόνο να βοηθήσουμε το, τον κλάδο, θα έλεγα, αλλά θα έλεγα πως εμείς εντός των κοινοτήτων αντιμετωπίζουμε τις καμήλες που αναφέρατε πριν ως προϊόν της διαδικασίας. Εργαζόμαστε λοιπόν επιτόπου στα δικαστήρια για τους ε, πολίτες ε, κάθε μέρα και στην διαδικασία αυτή συλλέγουμε πληροφορίες ε, και βλέπουμε πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί ίσως να βελτιωθεί. Αυτό το οποίο κάνει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου είναι κάποια έργα που αναλαμβάνει που δεν είναι τόσο ακαδημαϊκού χαρακτήρα, έχουν μια γεύση πρακτικής πτυχής, αφορούν κάποιες πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου, κάποιες από τις οποίες αναφέραμε ήδη, και ακριβώς συνεισφέρουμε με την πείρα των ανθρώπων που εργάζονται κάθε μέρα πάνω σε αυτό το θέμα, την πείρα των δικαστών και την πείρα των πανεπιστημιακών και μπορούμε έτσι να παρουσιάσουμε ένα προϊόν το οποίο δείχνει πώς μπορεί να βελτιωθεί ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το εάν τώρα θα τα ακούσετε αυτά ή όχι είναι οπωσδήποτε δική σας επιλογή ως νομοθετικό σώμα. Αλλά εμείς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε και έχοντας την εμπειρία του Ευρωβουλευτή θεωρώ πως η ανεξάρτητη αυτή δουλειά μπορεί καμιά φορά να βοηθήσει να ξεπεραστούν ε, διάφορες ε, στενοποίησεις στο πολιτικό σύστημα. Είμαστε λοιπόν διάφοροι νομικοί, ευρωπαϊκή νομική κοινότητα θα έλεγα, που είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας σε διάφορα ζητήματα. Αναφέρθηκε το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων, το οικογενειακό δίκαιο, όλα αυτά είναι τομείς ε, που μας απασχόλησαν. Είχαμε επαφές με πολλούς από εσάς. Είμαστε στην διάθεσή σας να βοηθήσουμε όσο εσείς θέλετε. Πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν θέλουν και οι συνάδελφοί να πούν κάτι, αλλιώς είμαστε στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε. Είναι μεγάλη τιμή και νιώθω μεγάλο προνόμιο που ξαναβρισκόμαστε εδώ και μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου. Θα ήθελα, συντομία, να επανέλθω σε αυτά που είπε η πρόεδρος Wallis για το τι ιδιαίτερα έχουν τα σχέδια του Ινστιτούτου μας και ποια είναι η προσεθέμενη αξία του έργου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι το εξή. Όλα τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου είναι το αποτέλεσμα μια συλλογική προσπάθειας ενός ε, μεγάλου φάσματος ε, νομικών και νομομαθών που έχουν ε, διαφορετική επαγγελματική πείρα, συμβολογράφοι, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί, δικαστές, νομομαθείς και νομικοί από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης και εκπρόσωποι διαφόρων νομικών παραδόσεων. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι γνωρίζετε τι έκανε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Είχαμε μια ομάδα εργασίας που απαρτιζόταν από δικαστές, ε, καθηγητές πανεπιστημίου και δικηγόρους ε, με πρόεδρο τον ε, Λόρδο Τόμας από την Ουαλία. Και δεν ήταν μόνο μια ομάδα εργασίας, ήταν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου που συνέβαλαν στο επώνυμα αυτό. Περίπου χίλια, χίλια φυσικά πρόσωπα και πολλοί παρατηρητές και άλλα Ινστιτούτα που προσέφεραν τις παρατηρήσεις τους σε διαβουλεύσεις που κράτησαν περίπου ένα χρόνο. Και η ομάδα εργασίας μας έλαβε υπόψη όλες τις πληροφορίες και τις προτάσεις και ανέλησε διεξοδικά και εξονυχιστικά όλα τα προ... όλα τα... όλες τις προτάσεις. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε και με φοιτητές διδακτορικού που είχαν την ευκαιρία και αυτοί να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και σχόλιά τους. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Ποιο, πώς διαμορφώνονται τα πονήματά μας. Επίσης, ε, είμαστε απόλυτα ανεξάρτητοι από τους ηθήνοντες πολιτικής και από ε, εκπροσώπους συμφερόντων. Έχουμε βέβαια εκπροσώπους ε, από διάφορους κλάδους για παράδειγμα, είχαμε την CCB στην ομάδα εργασία, τη CCJ, διάφορε ε, ενώσει και εκπροσώπου του. Αλλά όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι, ε, επειδή το έργο του ανεξάρτητα από την οργάνωση από την οποία προέρχονταν. Και ε, είδαμε τις αποφάσεις ε, των ε, ευρωπαϊκών οργάνων, τις θεωρούμε ως δεδομένες και όπως είπε η Νταϊάννα, εμείς επικεντρωνόμαστε σε τεχνικά θέματα, σε τεχνικές πτυχές και λέμε αν θέλετε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο πωλήσεων, πώς θα πρέπει να το διαμορφώσετε για να γίνει πιο εύχριστο στην πράξη και να εξυπηρετεί πραγματικά τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης, τρίτο και τελευταίο σχόλιο ανέκαθεν προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα χειροπιαστά, αυτά και άμεσης ε, χρήσης. Γιατί ε, μπορεί να σε ακαδημαϊκό, να ασχολείται με θεωρητικά θέματα, αλλά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Είναι υποχρεωμένο να υποβάλει έμπρακτε προτάσει και λύσει. Αλλιώ ε, δεν θα ήταν χρήσιμο το έργο μα. Και αυτό το λέμε σε όλε μα τι δηλώσει. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες ε, σε εσά και περιμένουμε ανυπόμονα τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το έργο μας και τι περιμένετε από μας και πώς κρίνετε τη μέχρι τώρα μεθοδολογία μας. Σας βοήθησε, μπορεί να είναι εύχρηστη και στο μέλλον, εξυπηρετεί την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, στο εκτελεστικό όργανο του Ινστιτούτου μας ε, εστιάζουμε στη συνεργασία των Ινστιτούτων, του Ινστιτούτου με άλλα ε, μη ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, οργανώσεις όπως η Unitral, αλλά δεδομένες της ιστορίας και του μοντέλου που χρησιμοποίησαμε, συνεργαζόμαστε στενά με το Αμερικανικό Ινστιτούτο και την ε, Αμερικανική Επιτροπή για νομικά θέματα των ΗΠΑ. Δεν είναι ότι θέλουμε να φέρουμε το αμερικανικό δίκαιο στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε να εμπνευστούμε απλώ από αυτού. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο είναι διαβόητο για τις ε, πρακτικές του που επηρεάζουν πολύ την ε, νομική πρακτική, τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Έχουν μοντέλα για τους νόμους. Συνεργάζεται με την Αμερικανική Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη. Ε, και σχεδιάζουν μοντέρνους νόμους που θα εφαρμοστούν από τις διάφορες πολιτείες. Δηλαδή, ε, εναρμόνιση ή ενοποίηση από κάτω προς τα πάνω. Κοιτάμε αυτά τα δύο Ινστιτούτα τι κάνουν μαζί και αυτό μας βοηθάει γιατί ε, όπως και εμείς στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε την επικουρικότητα ως έμπνευση, έτσι και αυτοί χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο. Ε, ίσως αυτό σας φαίνεται αντίφαση, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Αμερικανική Επιτροπή ε, πρόσφατα ε, ε, έκανε ένα νόμο για την πρόσβαση σε στοιχεία του εταιρικού εταιριών ε, που ασχολούνται με ψηφιακά θέματα. Ε, επίσης οι Αμερικάνοι συνεργάζονται με τους Καναδούς για αυτά τα θέματα. Συνεργαζόμαστε για να δούμε αν αυτός ο νόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να είναι ένα ευρωπαϊκό μέτρο, θα μπορούσε να είναι ένας νόμος μοντέλο που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε στα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και με αυτούς. Ε, συνεργαζόμαστε με την Ασιτράλ και την Unidra. Προσπαθούμε να πάρουμε ιδέες από οποιονδήποτε. Και όπως ακούσαμε και από τον Επίτροπο, ε, να εμπνευστούμε για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν εκτός της Ευρώπης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και η Ευρώπη είναι τμήμα ενός ευρύτερου κόσμου. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό δουλεύοντας ανεξάρτητα ε, με σκοπό το τι πρέπει να γίνει στην πράξη. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ε, αν μας δώσετε ιδέες θα τις ακούσουμε με μεγάλη χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ και τους τρεις που μας κάνετε αυτές τις παρουσιάσεις για το δυναμικό του Ινστιτούτου σας. Και εγώ προσωπικά, από τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση, έχω να μαρτυρήσω ότι οι εμπειρογνώμονες που έχετε, ε, ο κόσμος που έχετε, ε, έχει ωραίες ιδέες. Ε, ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να χαιρετήσω την πρόεδρο της οργάνωσής σας, την οποία εμπιστεύομαι απόλυτα, την Ταϊάννα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που δεν τους ξέρω. Ε, και επιπλέον δεν, έχω την, δεν είχα την ίδια καριέρα. Το ερώτημά μου είναι το εξής το Ινστιτούτο σας θα συνεισφέρει στην απλούτε, απλούστευση του δικαίου που παράγουν τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δουλεύετε δηλαδή υπέρ της απλούστευσης της ε, ευρωπαϊκής ε, δικαιοσύνης, του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα πρέπει το παραγόμενο δικαίο, δίκαιο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι κατανοητό και άμεσα χρήσιμο για τους πολίτες. σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν να επιλύσουν, σε σχέση με, την, με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κτλ. Να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και θα απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Σβιεύκα. Ευχαριστώ. Αισθάνομαι απεριόριστη χαρά που ξαναβλέπω την Ταϊάννα στη συνεδρίαση της Νομικής Επιτροπής, παρόλο που τώρα έχει πολύ διαφορετική ιδιότητα αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την ε, επαφή, γιατί για χρόνια ολόκληρα είχαμε συνεργαστεί και αυτή η παλιά συνεργασία θα μας ε, χρησιμεύσει και στο μέλλον που θα αναπτύξουμε ενός νέου είδους συνεργασίας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σχέδια και θέματα που απασχολούν το Ινστιτούτο. Ξέρω ότι ε, επεξεργάσετε ένα όραμα προκειμένου να βοηθήσετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να υλοποιήσουν το καθήκον τους και την αποστολή τους, να εκπονήσουν σωστές νομοθετικές διατάξεις και σωστό καλό δίκαιο. Το θέμα της συνεργασίας ε, με ενδιαφέρει, της ε, δικαστικής συνεργασίας για το σχέδιο που σας απασχολεί που έχει τίτλο «Από τις διασυνοριακές αρχές σε ευρωπαϊκούς κανόνες για αστικές υποθέσεις». Το σχέδιο αυτό κάνει μία ανάλυση της εναρμόνισης των διασυνοριακών αστικών διαδικασιών και δικών. Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στο, στην αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε όλες τις ε, χώρες μέλη, άσχετα από το που εκδόθηκε σχετική, η σχετική δικαστική απόφαση. Τώρα, σε σχέση με το δικό σας σχέδιο, θα περιμένουμε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κάποιες αλλαγές ε, στη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Ή μήπως βλέπετε σε αυτό το στάδιο αναγκαία ήδη την εναρμόνιση. Ή μήπως προτιμάτε να εμείνουμε στις υφιστάμενες αρχές ε, ε, δικαστικής συνεργασίας που στηρίζεται, όπως είπα, στην αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, είπε σε μία δήλωσή του ότι είναι σημαντικό να αφήσουμε κάποια θέματα στην εθνική αρμοδιότητα και στην ε, συνεργασία μεταξύ των κρατών μέλων. Πολλά ε, επαφίονται σε αυτό. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση ή για μια προσπάθεια ανάλυσης της μέχρι τώρα κατάστασης και τι λύσεις ε, ή τι μοντέλο κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο αποτελεσματικό. Η κυρία Ρέζα. Thank you very much. Uh, I'm very glad that... Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερω που είχατε την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου και εμείς ως μέλη της Νομικής Επιτροπής στηριζόμαστε στην πυρογνωσία και των πανεπιστημιακών αλλά και νομικών και δικηγόρων για να βοηθούμε στο έργο μας να υποβάλουμε σωστές νομοθετικές προτάσεις. Μια και αναφερθήκατε στο θέμα της ψηφιοποίησης και τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το διαδίκτυο, ε, θα ήθελα να πω ότι από τη συνθήκη της, Ευρω... της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά σχέδια εναρμόνισης στο τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Και τώρα αρχίζουμε και την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το copyright. Θεωρείται ότι η εισαγωγή ενός τίτλου copyright πανευρωπαϊκού θα μας επιτρέψει να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε εξαιτίας της διασυνοριακής πρόσβασης σε διάφορα έργα και πιστεύετε ότι έτσι θα ενισχυθεί και η διαφάνεια του δικαίου για τους καταναλωτές. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Πρόεδρο την κυρία Γόλης και στους συναδέλφους της ε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Διαλέξτε εσείς με ποια σειρά θα απαντήσετε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Κύριε Καβαντά, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, ένας από τους λόγους ύπαρξης του Ινστιτούτου μας είναι να βελτιώσουμε την ενωσιακή νομοθεσία. Και αυτή τη λειτουργία και την αποστολή έχει και το αντίστοιχο Αμερικανικό Ινστιτούτο Δικαίου. Τον ίδιο στόχο έχουμε και εμείς να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέλουμε να γίνει πιο προσιτό, σίγουρα, το δίκαιο αυτό. Και μάλιστα, ε, όσο ήμουν ευρωβουλευτής, ασχολήθηκα με κάποιες ε, ε, επιτομές που συντάξαμε για τους πολίτες για να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με την κοινωτική νομοθεσία. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι προσιτή ενωσιακή νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και όπως είπε και η συνάδελφος, το έργο μας δεν είναι άσκηση κριτικής. Απλώς θέτουμε επιτάπητος ε, όλους τους ε, κανόνες που μπορούν να είναι χρήσιμοι. Εμείς δεν επικρίνουμε κανένα, δεν ασκούμε κριτική για τις προτάσεις, αλλά απλώς δίνουμε κάποιες χειροπιαστές ε, δυνατότητες για να βελτιωθεί η κοινοτική νομοθεσία στους τομείς που εξετάζουμε. Και ευελπιστώ ότι έχουμε ως προς την άποψη αυτή κοινό στόχο. Κύριε Σβιεύκα, ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνατε για τα σχέδια που αφορούν ε, τη διαδικασία στις αστικές υποθέσεις και τη δυνατότητα μιας ευρωπαϊκής διαδικασίας. Με ενδιαφέρει το θέμα αυτό, το θεωρώ συναρπαστικό από πολλούς και διάφορους ε, λόγους και απόψεις και είχαμε και στο παρελθόν κοινό ενδιαφέρον ε, μαζί με τη UNIDUA εκπονώ αυτό το σχέδιο. Η UNIDUA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, μία από τις οργανώσεις που είναι μέλη. Και το έχουμε μία δέσμη κανόνων για τις Ευρώπης, για τις αστικές διαδικασίες, για τις διαδικασίες αστικές υποθέσεις, ε, ίσως έχει νόημα, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουμε σύνη στις ένομες τάξεις μας και στα δικαϊκά μας συστήματα. Υπάρχουν όμως και κάποιες τεχνικές ε, λεπτομέρειες που στηρίζονται στον κανονισμό Βρυξέλλες 1 και υπάρχουν και τεχνικές λεπτομέρειες που οφείλονται στις διαφορές των ε, δικαιικών μας συστημάτων. Χρειάζεται και μια τεχνική προεργασία ώστε να έχουμε καλύτερη διαπαφή των διαφόρων νομικών συστημάτων και τάξεων. Αυτή τη στιγμή Έχουμε τέσσερις ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από πολλούς ε, επαγγελματίες ε, σε θέματα νομικά και έχουμε στενές και τακτικές επαφές με τον πρόεδρό σας και προτείνω στη συνέχεια, ίσως τον Απρίλιο θα είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχετε με μέλη αυτών των ομάδων εργασίας, προκειμένου να γίνουν παρουσιάσεις και να ενημερωθείτε για το έργο αυτών των ομάδων. Πάντως, αν καταλήξουμε σε κάποιες ευρωπαϊκές αρχές για τις αστικές δίκες, θα χρησιμοποιηθούν και θα έχουν και πολιτική βαρύτητα, όχι μόνο εδώ, αλλά και στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό το επιπλέον δέλερ θα δημιουργήσει και η συμμετοχή της UNIDWA. Και πιστεύω ότι έτσι θα, δούμε πρόοδο στην ευρωπαϊκή διαδικασία για τις αστικές υποθέσεις. Πάντως θα επανέλθουμε για να σα δώσουμε πιο πολλές λεπτομέρειες για τα επιμέρους αυτά σχέδια που επεξεργαζόμαστε. Ευχαριστώ και για την ερώτηση για την ψηφιοποίηση, για το δίκαιο που έχει σχέση με τα ψηφιακά θέματα και το νέο δίκαιο για το copyright. Ήδη έχουμε μια ολιγομελή ομάδα εισηγητών που εκπώνησαν μια αρχική έκθεση μετά τις περσινές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για το θέμα αυτό και αν έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε και εμείς στο έργο σας θα το κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Αυτά από μέρος μου. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να συμπληρώσουν αν έχουν κάτι. Να επανέλθω λίγο στις αρχές της δουλειάς μας. Μας ρωτήσατε αν πιστεύουμε πως ε, ο ευρωπαϊκός τίτλος copyright είναι η σωστή ε, Δεν μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή γιατί μόλις ξεκίνησε η δουλειά. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας ε, που θα ξεκινήσει τα μέλη του Ινστιτούτου θα συνεισφέρουν. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας πούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το συναρπαστικό στη δουλειά μας. Έτσι δουλεύουμε. Όπως ξέρετε, οτιδήποτε σχετίζεται με το ίντερνετ εξορισμού δεν έχει σύνορα, οπότε οποιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται στην Ευρώπη πρέπει να γίνει δεκτή παγκοσμίω. Γι' αυτό ακριβώς η συνεργασία νομίζω με το αντίστοιχο Αμερικανικό Ινστιτούτο και άλλους οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι απολύτως απαραίτητη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως τα δεδομένα ρέουν και μπορεί κανείς να τα κατεβάσει οπουδήποτε. Μπορεί μια χώρα να αποκοπεί από το διαδίκτυο, αλλά μετά Βεβαίω ε, κάτι τέτοιο αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν προγράμματα που παρακάμπτουν ε, τα πάντα. Ε, ξέρω πώς γίνεται κατάχρηση, αλλά η τεχνολογία υπάρχει. Οπότε, πούμε, δεν, δεν έχουμε κάποια θέση αυτή τη στιγμή. Καλή ιδέα που προτείνεται, αλλά εμείς δεν θα την προτείναμε αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερη έρευνα και βεβαίως να δούμε και εκτός Ευρώπης, αν ε, θα μας ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλη μια ερώτηση, ο κ. Μπούντα, αν μας επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γουόλης. Η δραστηριότητά σας είναι πάρα πολύ σημαντική Γιατί βεβαίως ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε κάποιες απόλυτες αλήθειες. Έχω κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αύριο θα συζητήσουμε ένα θέμα, σας έχει απασχολήσει καθόλου το ζήτημα αυτό των μικροδιαφορών και της ευρωπαϊκής ε, εντολής ε, πληρωμής. Θα συζητάμε αυτά και κοιτώντας τις τροπολογίες δεν ξέρω, κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να φύγουν, να, να φύγει αυτή η διαδικασία, άλλοι τη δέχονται. Το ζήτημα αλλού είναι το ποσό πάνω από το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία. Ότι άλλοι λένε ότι θα πρέπει να ανέβει το κατόφλι για να είναι προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Έχετε κάνει κάποια μελέτη, τι άποψη έχετε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω πως πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Η απάντησή μου είναι παρόμοια με αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Ε, δεν μας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα. Έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν ε, είναι σωστό να πω πως είναι η άποψη του Ινστιτούτου αλλά μπορώ να πω πως στο μέλλον και διστάζαμε κάπως είπα πως είμαστε μια κάπως ένας κάπως νέος οργανισμός και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η νέα Κομισιόν και πως στο μέλλον μπορούμε να βοηθήσουμε και πρέπει να πω, θα έπρεπε να έχω πει πριν, πως ε, η κυρία Σβίφκα το είπε άλλωστε, πως η Κομισιόν παρακολουθεί την διαδικασία, είναι στην, ε, στις ε, συνεδριάσεις μας και θα δούμε τι θα προκύψει. Αλλιώς θα μπορούσα να σας δώσω μία προσωπική απάντηση, αλλά δεν είναι απάντηση του Ινστιτούτου. Αυτά και δεν μπορώ να σας βοηθήσω αυτή τη στιγμή για αυτούς, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρξουν και κάποια πράγματα. Λοιπόν, τελείωσαν νομίζω οι ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την πρόεδρο ε, να ευχαριστήσω την πρόεδρο Γόλης και τους καθηγητές που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα και είμαι σίγουρος πως δεν θα είναι τελευταία φορά. Ε, we continue with ε, number eight. Με το σημείο 8 της ημερήσης διάταξής μας έχουμε μία ακόμη παρουσίαση για σήμερα. Έχουμε την χαρά να υποδεχθούμε εδώ τον Λόρδο Watch ε, από πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Ουαλίας και Σκοτίας και ε, ως πρώην και έμπειρος δικαστής ε, θα μας ενημερώσει για θέματα που μας ενδιαφέρουν, ιδιαίτερα εταιρικό δίκαιο, αφαιρικιότητα, πνευματικά δικαιώματα, Εγγύησης και ούτω καθεξής. Αλλά σήμερα θα μας μιλήσει ειδικά για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων. Ο Λούτζι Μπερλιγκουέρ ήταν ο πρώτος πρόεδρος αυτού του δικτύου, ένα πρώην επιφανέστατο μέλος της Νομικής Επιτροπής. Λόρδε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή. Ελπίζω οι ερωτήσεις να μην επεκταθούν σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Εγώ σήμερα θα ήθελα κάτι άλλο να σας εξηγήσω. Να σας εξηγήσω συντομία τι εστί Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων. Τι κάνει ήδη τώρα και τι προσφέρει για το μέλλον. Καταρχήν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Δικαστικών Συμβολίων είναι ένα θεσμικό δίκτυο που απαρτίζεται από 20 μέλη δικαστικά συμβούλια, από 17 χώρες μέλη και 15 παρατηρητές από χώρες μέλη που δεν έχουν δικαστικά συμβούλια, δεν έχουν αυτό το θεσμό στην ενωμή της τάξη. 8 ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και 7 ε, είναι παρατηρητές από υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό καταρχήν να ξέρουμε τι είναι και τι κάνει ένα δικαστικό συμβούλιο γιατί αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της συνταγματικής μας ένωμης τάξης. Ένα τέτοιο δικαστικό συμβούλιο προσφέρει την προστασία που χρειάζεται κάθε δημοκρατικό κράτος για την ανεξαρτησία του δικαστικού της κλάδου, της δικαστικής εξουσίας και την προαγωγή του κράτους δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη αν δεν έχουμε στην ένωμη μας τάξη και ένα δικαστικό συμβούλιο. Ένα συμβούλιο ε, για τη δικαστική εξουσία. Αλλά απλώ τέτοιου είδου δικαστικά συμβούλια αποτελούν το πιο αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μοντέλο ή λύση για να διαχωρίσουν την τρίτη εξουσία, τη δικαστική, και να τη διακρίνουν από, τις ε, δύο άλλες, ε, από τους δύο άλλους ε, εξουσίας, την ομοθετική και την εκτελεστική. Ουσιαστικά το Δικαστικό Συμβουλίο είναι ένας προφυλακτήρας και επιτρέπει το δικαστικό και δικαιωτικό σύστημα να τη χάνει ανεξάρτητης διαχείρισης, ανεξάρτητης από τα άλλα θεσμικά όργανα που μερικές φορές μάλιστα θα κληθεί να, να κρίνει και σε διάφορες σχετικές υποθέσεις. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιτρέπει στα ε, δικαστικά συμβούλια των χωρών μελών να ξεκινήσουν διάλογο για να βελτιώσουν τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους και να προωθήσουν ταυτόχρονα βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουν οι δικαστικές ε, ε, εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουν και να απονείμουν ποιοτική, αποτελεσματική και έγκαιρη δικαιοσύνη. Κάτι που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μυστικό ότι η καιροί είναι χαλεπή για πολλές δικαστικές τάξεις και ακόμη και για χώρες μέλη. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων συνεργάζονται για να βελτιώσουν όλα τα δικαιικά και δικαστικά συστήματα, γιατί κανένα δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο. Το Ευρωπαϊκό Αυτό Δικτύο διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και έτσι σταδιακά, σιγά σιγά θα καταλήξουμε ενδεχομένω σε μια ευρωπαϊκή δικαστική και νομική παιδεία, κουλτούρα. Γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε και να προωθήσουμε κοινέ αρχές, αξίες και πρακτικές. Και μάλιστα ναι, οι δραστηριότητες μας ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ δικαστών και του δικαστικού κλάδου γενικώ. Και μάλιστα τα, οι ομάδε μα έχουν καταλήξει σε κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ σε τομεί όπω είναι η διαντολογία, η δικαστική, πρόθεση, ε, η διορισμό και προαγωγή των δικαστών, αξιολόγηση και μονιμότητα των δικαστών, εμπιστοσύνη του κοινού στους δικαστές και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών. Μάλιστα έχουμε φέτος ένα σχέδιο για προδιαγραφές για την δικαστική πειθαρχία. Πολύ σημαντικό θέμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες μέλη. Και για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων ασχολείται και με κατάρτιση δικαστών και συνεργαζόμαστε ενεργά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κατάρτιση των Δικαστών. Πρόσφατα ε, έγινα πρόεδρος αυτού του δικτύου και όχι μόνο θέλω να θεσπιστούν πρότυπα, αλλά θέλω στην επόμενη φάση ανάπτυξη του δικτύου να εφαρμοστούν αυτά τα πρότυπα. Και ελπίζω ότι στο μέλλον θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών και των κατευθυντηρίων γραμμών και θα βελτιωθεί έτσι τα δικαστικά συστήματα, ε, μια και θα υπάρξει συμμόρφωση με τα πρότυπα τα τελευταία χρόνια ε, υπάρχει ένα σύστημα όπου τα, μέλη, τα συμβούλια που είναι μέλη και οι παρατηρητές μπορούν ενεργά να αναζητήσουν βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων όταν έχουν ειδικά, ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, αυτό το χρησιμοποίησαν συμβούλια στη Σλοβακία, Βοσνία Ερσεγοβίνη και πρόσφατα στην Αλβανία. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο αυτό εμπλέκεται ενεργά στην δεύτερη χρονιά ενός φιλόδοξου προγράμματος που θέλει να αναπτύξει και να εφαρμόσει δείκτες για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας του δικαστικού κλάδου στα κράτη-μέλη. Δημιουργούμε μικρές ομάδες διαλόγου με τέσσερα μέλη ή παρατηρητές με σκοπό να βρεθούν λύσεις για την βελτίωση κάθε δικαστικού συστήματος ειδικά στους τομείς που έχει και παρουσιάζει προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ φιλοδόξο γιατί τα δικαστικά συστήματα και τα δικαστικά συμβούλια δεν επιθυμούν πάντα να διερευνήσουν τους προβληματικούς τομείς τους. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προωθεί επίσης ε, ε, την έγκαιρη και αποτελεσματική δικαιοσύνη. Η καθυστέρηση είναι ο εχθρός της δικαιοσύνης και η συσσόρευση υποθέσεων είναι πολύ προβληματικό θέμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, κάνει περιφερειακά σεμινάρια με σκοπό να βρεθούν λύσεις σε αυτά τα επίγοντα προβλήματα. Τα πρόσφατα χρόνια το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, ενεργά ε, δραστηριοποιήθηκε και συνεργάστηκε με την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης για τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη. Θέλουμε ε, να μετρήσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και πιστεύουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ε, βοηθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και το δίκτυο υποστήριξε τις προσπάθειες της Κομισιόν για τον ε, πίνακα αποτελεσμάτων. Αν λειτουργούν τα δικαστικά συστήματα, μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτε να ασκήσουν τα δικαιώματά του. Η ανεξαρτησία και η εργοδοσία τη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική για να γίνουν τα παραπάνω. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η, η... σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου θα δεν θα γίνει και οι πολίτες δεν θα έχουν τα απαραίτητα ένδικα μέσα ε, που προβλέπει η χάρτα. Στο μέλλον, το όραμά μας είναι να υπάρξει μια ευρύτερη κατανόηση της σημασίας και της σωστής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι δικαστές όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη για πραγματική ε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πραγματική λογοδοσία των δικαστικών συστημάτων, ε, η έλλειψη διαφάνειας που παρουσιάζουν πολλά συστήματα και η υποχρηματοδότηση είναι κάτι που είναι παράδεκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπαίδευση και του κοινού αλλά και των δικαστών είναι κλειδί για να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαστικά συστήματα θα υπηρετούν καλύτερα τους πολίτες για τους οποίους, είναι, για τους οποίους υπάρχουν. Ως πρόεδρος, κατά διάρκεια της αιτίας μου πρόεδρος του δικτύου, θέλω να βελτιώσουμε την συνεργασία του δικτύου με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω ότι οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι δικαστές και τα συμβούλια, τα δικαστικά, όλα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση ως το μόνο πραγματικά θεσμοθετημένο δίκτυο που ασχολείται για τη δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει το δίκτυό μας να είναι προπομπό για τη βελτίωση των προτύπων, να εντοπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συμβούλια σε όλη την Ευρώπη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δικαστικά συστήματα και να προωθήσουμε πραγματικέ και αποτελεσματικέ λύσει. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει τη διαφορά βοηθώντας την ε, Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο και χάρη στην περαιτέρω συνεργασία μας θα, θα δημιουργήσουμε ακόμα πιο ποιοτικά δικαστικά συστήματα. Το δίκτυο και τα μέλη του μπορούν να προσφέρουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ένα όραμα από τη σκοπιά της δικαιοσύνης για νομικά και άλλα θέματα που παρεμποδίζουν την ε, απόδοση, την απονομή της δικαιοσύνης. Και Γι' αυτό ακριβώς ε, ε, παρακολουθούμε τη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι κυρίως για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις για τα θέματα που μίλησα, για την αφαιρεγγιότητα, για το copyright και για όλες τις άλλες πτυχέ θα μπορούσα να μιλήσω, για τι οποίε έχω ασχοληθεί στο παρελθόν στην καριέρα μου, που αναφέρατε εσεί, Πρόεδρε, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε τον χρόνο. Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα, που μα δείχνετε όχι μόνο τη σημασία τη δουλειά σα, αλλά και το δυναμικό που έχει και τι μπορείτε να προσφέρετε σε αυτό το Ινστιτούτο. Με χαρά βλέπω ότι μπορείτε να καλύψετε πολλούς τομείς δικαίου που μας απασχολούν και εμάς, που μας ενδιαφέρουν και εμάς. Αλλά παρακαλώ του ευρωβουλευτέ να μην κάνουν τέτοιε ερωτήσει, αλλά να επικεντρωθούν στην ουσία Τη παρουσίαση του Λόρδου μέλους της Νομικής Επιτροπής του Βουλή των Λόρδων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ερώτηση. Απλά θέλω να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζω εδώ τον Λόρδο σήμερα. Θα θυμάστε μάλιστα πως την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν όπου νομίζω κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά και εκεί. Ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως ε, η Επιτροπή μας οπωσδήποτε θα συνεργαστεί πλήρως μαζί σας και θα είμαστε αξιόπιστος εταίρος και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε σήμερα εδώ. Άλλες ερωτήσεις από τους βουλευτές. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Μαρίνιου Πίντου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια γνήσια μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη καλύτερα ένα εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς είναι δυνατόν να έχουμε κάτι τέτοιο και να το προσαρμόσουμε σε ανάγκες της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, της οικονομίας και της ηθαγένειας. Υπάρχουν τόσο διαφορετικές λύσεις εξαιτία των διαφορών των εθνικών νομοτάξεων. Οπότε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη δικαιοσύνη. Ποιος είναι ο ιδανικός ε, δικαστής και πώς, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος απονομής ε, της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι ένας πραγματικός δικαστής ένας νέος 25, 26, 27 ετών που καταρτίστηκε σε μια επαγγελματική σχολή δικαστών. Αρκεί αυτό ή μήπως χρειάζεται και εμπειρία ζωής, μια οριμότητα και κοινή λογική, κοινό νους που τη δίνει πολλές φορές μια επαγγελματική προηγούμενη πείρα και όχι απλώς μια φίτηση σε μια σχολή δικαστών. Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση της δικαιοσύνης σε πολλές χώρες, όπως στην Πορτογαλία, είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό της εθνικής κυριαρχίας. Και παρόλα αυτά, οι δικαστές και οι εισαγγελεί είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα, σαν να ήταν ε, τυχαίοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και μάλιστα ε, μπορούν να ασκούν και το δικαίωμα τη απεργία. Κάτι τέτοιο είναι συμβατό με την ιδέα της δικαιοσύνη που θα πρέπει να είναι υπεράνω τέτοιων ε, πολιτικών ή άλλων συμφερόντων που υπάρχουν μερικές φορές και χαρακτηρίζουν τη συνδικαλιστική δράση. Τέλος. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση, τι εχέγγυα μπορούμε να θεσπίσουμε, ώστε ε, να έχουμε μια πραγματική διάκριση των εξουσιών. Γιατί εγώ είχα εμπειρία ως δικηγόρος και ήμουν και πρόεδρος και του Πορτογαλικού Δικαστικού Συλλόγου, Δικηγορικού Συλλόγου, συγγνώμη, ε, και έχω την αίσθηση ότι σε περισσότερες, περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα εθνικά κοινοβούλια δεν ενδιαφέρονται για πραγματική διάκριση μεταξύ της δικαιοσύνης και της πολιτικής. Και έχουμε όλο και περισσότερα φαινόμενα πολιτικοποίησης της δικαιοσύνης. Και αυτό το βλέπουμε στην πατρίδα μου, την Πορτογαλία, αλλά και ολού. Ή έχουμε και το αντίστροφο φαινόμενο δικαιοποίησης της πολιτικής. Δηλαδή, η δικαιοσύνη να εξυπηρετεί κομματικά ή πολιτικά συμφέροντα κάτι που κανονικά δεν επιτρέπεται. Τι λύσεις μπορείτε να προσφέρετε για το πρόβλημα αυτό, αν φυσικά το κρίνετε ως πρόβλημα, όπως ε, εγώ πιστεύω. Ε, Ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, οπότε έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Νομίζω πως οι απαντήσεις ε, θα χρειαζόταν δυόμιση ώρες. Οπότε θα είμαι σύντομο τώρα πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την ε, δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα σταδιακά. Δεν γίνονται αυτά σε μία μέρα. Αλλά με τη συνεργασία της δικαιοσύνης διαφόρων χωρών ε, και με το Συμβούλιο μπορούν νομίζω να ε, διδαχτούν οι χώρες η μία από την άλλη και να δουν τα καλά του κάθε συστήματος. Σημαντικό αυτό το οποίο είπατε ότι δηλαδή πρέπει να δούμε και την εξέλιξη της οικονομίας. Αυτό το οποίο λέω εγώ πάντα και νομίζω είναι σημαντικό είναι πως καμία οικονομική ένωση και καμία οικονομία δεν μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς ένα επιτυχές σύστημα δικαιοσύνης ε, στο οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και οι πολίτες. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η δικαιοσύνη για μια επιτυχημένη οικονομία. Και άρα το οφείλουμε στους πολίτες μας να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης σε κάθε κράτος μέλος, αλλιώς η οικονομία της Ένωσης θα υποφέρει. Μετά αναφερθήκατε στην ηλικία των δικαστών. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος στην Ευρώπη θεωρεί πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των συστημάτων ε, της Ευρώπης, ε, του αστικού δικαίου και αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου και θεωρούν πως δεν υπάρχει συνεννόηση. Λάθος. Κάθε σύστημα δικαιοσύνης έχει τον ίδιο στόχο να προσφέρει δικαιοσύνη σε ο κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Είτε μιλάμε για δικαιοσύνη στον τομέα τον διοικητικό, τον αστικό, τον ποινικό, οικογενειακό κτλ. Και διαφέρουν ελαφρώς οι ρίζες για την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά γεγονός είναι πως υπάρχει περιθώριο για να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος με διαφορετικούς τρόπους. Και έχω μελετήσει συστήματα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο παρόμοια είναι διαφορετικά συστήματα δικαιοσύνης όταν αφαιρέσουμε όλη την επιφάνεια στην οποία στέκονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Οπότε δεν έχω κάποια αμφιβολία για το ότι μπορεί να υπάρχουν νέοι δικαστές, εκπαιδευμένοι, πετυχημένοι. Στην ηλικία μου όλοι οι δικαστές είναι ηλικιωμένοι, σαν και εμένα, ίσως να μην είναι πολύ καλή ιδέα. Ε, θα ήταν να αλλάξει. Και ε, θα είμαι σύντομος ε, κύριε Πρόεδρε, μετά ερχόμαστε στο ζήτημα των ε, ενώσεων των δικαστών. Σε κάποιες χώρες είναι ισχυρές αυτές οι ενώσεις, αλλά ένα θεσμικό δίκτυο όπως το δικό μας υπάρχει ακριβώς για να διασφαλίσει πως υπάρχει η απαραίτητη ανεξαρτησία και λογοδοσία της δικαιοσύνης προς όφελος των πολιτών. Βεβαίως πρέπει να μπορούν και οι δικαστές να αναφέρουν τα αιτήματά τους, αλλά απέχουμε πολύ από αυτό. Εμείς εξετάζουμε την δομή του συστήματος που υπηρετεί την χώρα και το κράτος. Και πραγματικά εκπροσωπούμε, όπως είπα, την ε, τρίτη εξουσία, όπως ε, ανέφερα. Συνολικά, λοιπόν, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τα συστήματα δικαιοσύνης ε, στην Ευρώπη. Θεωρώ πως θα βελτιωθούν και θα υπάρξει και αμοιβαία εμπιστοσύνη εάν συνεργαστούμε με τον τρόπο που προτείνει το δίκτυό μας. Οπότε είμαι σίγουρος πως όσο περνά ο καιρός τα συστήματά μας θα γίνονται καλύτερα και θα υπάρχει και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο στόχος μου ως ε, πρόεδρος του δικτύου. Σας ευχαριστούμε κύριε Δικαστά. Να αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που μας ε, τιμήσατε με την ε, παρουσία σας και είμαι σίγουρος πως ε, θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του δικτύου στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. the following point... Το επόμενο σημείο είναι και των θυρών, οπότε θα παρακαλέσω όσους δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη συνεδρία κλεισμένων των θυρών να φύγουν. Ευχαριστώ.